Uh, good morning, good afternoon everybody. Βέβαια δεν τα κατάφερνα αυτό τελευταία, αλλά πρέπει να αρχίσουμε τη συνεδρίση, με συγχωρείτε. Αλλά είχα μια συνάντηση με τον πρόεδρο Σούλτ, δεν μπορούσα να έρθω νωρίτερα. Να αρχίσουμε με την έγκριση της μερίσιας διάταξης υπάρχει μία αλλαγή. Ένα αίτημα, από τον κύριο Ότσικ Βλάσεκ που είναι ο εισηγητής μας για τις νέες προτάσεις της Κομισιόν. για το μέσο διευκόλυνσης της απορρόφησης πόρων των χωρών που αντιμετωπίζουν χρηματοπιστωτικές δυσχέρειες και θα ήθελε να δεχθείτε να το συζητήσουμε ως πρώτο θέμα τώρα αντί για αύριο το πρωί στις 9 γιατί αύριο ο κύριος Βλάσεκ πρέπει να πάει στην Πράγα. Οπότε τα 6 και 7 θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε αύριο πριν την ψηφοφορία που θα αρχίσει στις 10.30. Οι εισηγητές έχουν ενημερωθεί. Εντάξει. Ωραία, γίνεται δεχτή αυτή η αλλαγή στην ημερήσια διάταξη και οι χρόνοι που προβλέπονται για τη συζήτηση είναι βεβαίως ενδεικτικοί. Το... Η συνεδρία μεταδίδεται μέσω web streaming, έχουμε διερμηνία για... σε 12 γλώσσες. Και αυτά όσον αφορά την έγκριση της ημερήσια διάταξης. Μπορεί να εγκριθεί λοιπόν η ημερήσια διάταξη αλλά η Μαρή Τερέ Σμιθ θέλει να πάρει το λόγο. Είμαι σκιώδης για την ε, εδαφική συνεργασία που ήταν σήμερα και αύριο θα με απούσα στην αρχή της ε, συνεδρίασης. Γιατί έχω μια σημαντική συνάντηση αύριο πρωί-πρωί στην ε, Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10-10.30 θα είμαι παρούσα. Πρόεδρος. Αυτό εξαρτάται και από το πώς θα προχωρήσει η συζήτηση. Αν είστε στην αίθουσα θα δούμε εάν μπορέσουμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό για τους ομίλους εδαφικής συνεργασίας σήμερα. Μα είπατε τα 6 και 7 θα είναι πριν την ψηφοφορία. Πριν την ψηφοφορία μεταξύ 9 και 10 και μισή. Αλλά δεν θα είστε. Δεν θα είστε η κυρία Σάντσος, μα θα γυρίσω γύρω στις 10.30. Ε, σκόπευα να επιστρέψω για τις ψηφοφορίες που νόμιζα πως ήταν σήμερα το απόγευμα. Το Αλλά νόμιζα πως ήταν και σήμερα το απόγευμα το θέμα μου. Πρόεδρος. Θα προσπαθήσουμε να το συζητήσουμε σήμερα. Μήπως μπορείτε να μιλήσετε στον κύριο Μποστινάρου. Μήπως μπορείτε να κάνετε κάποια εναλλαγή. Θα επανέλθουμε στη μέση διάταξη αν θέλετε να το συζητήσετε. Θα εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη όταν θα την εγκρίνουμε. Να περάσουμε λοιπόν τώρα στο σημείο 2. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Θα σας ενημερώσω αύριο για τις ε, αποφάσεις των συντονιστών. Και τώρα να περάσουμε στο σημείο 9 όπως είπαμε. Και δίνω το λόγο στον Όλζη Βλάσα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Βάλτε τα ακουστικά σας, θα μιλήσω τσέχικα. Πρόεδρος, μήπως είναι καλύτερα να ακούσετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σε βοηθήσει. Παρακαλώ η Επιτροπή να μας κάνει την παρουσίαση του θέματος. Και μετά θα ακούσουμε τον εισηγητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με χαρά είμαι στη συνεδρίαση της Ρέτζη. Έχω να έρθω δύο χρόνια. Στην τελευταία συνεδρίαση που ήμουν είπα ότι ήθελα να ξανάρθω και σήμερα ξανά ήρθα. Να σας παρουσιάσω λοιπόν τον τρυπημένη πρόταση για τον κανονισμό των διαθροτικών ταμείων. Η πρόταση αυτή ενεκρίθη από την Επιτροπή την 21η Μαΐου. Είναι αντίδραση στην οικονομική κρίση. Ο κανονισμός άλλαξε για να εισαχθεί το λεγόμενο topping up, συμπληρωματική χρηματοδότηση. Δύο στοιχεία. Είναι αύξηση κατά 10% της συγχρηματοδότησης, του ποσοστού χρηματοδότησης. Και επίσης έχουμε μια αλλαγή που στοχεύει ε, να ε, χρηματοδοτηθούν περισσότερο η Ρουμανία και η Σλοβακία. Οι προτάσεις μας στοχεύουν να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν την εφαρμογή των ε, διαρθρωτικών ταμείων. Θα επανέλθω και στα δύο στοιχεία που περιέχει λοιπόν αυτή η πρόταση τροποποίησης. Να πω δύο λόγια για το λεγόμενο topping up. Αυτό επιτρέπει οι χώρες προγράμματος, που είναι τρεις η εξή. Η Ελλάδα. Η Κύπρος πρόσφατα ζήτησε να ενταχθεί, αλλά προς το παρόν είναι Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία μέχρι τέλους του χρόνου. Ε, αλλά ε, έχει όπως είπα ζητήσει και η Κύπρος topping up στα πλαίσια του παρόντος κανονισμού. Το topping up λύγει ε, τέλος τρέχοντος έτους και θα ήταν άτοπο να μην επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτή η δυνατότητα μέχρι το τέλος αυτής της περίοδος προγραμματισμού. Έτσι θα είχαμε τη δυνατότητα να γίνουν νωρίτερα πληρωμές προς τις χώρες προγράμματος για την Ελλάδα. Αυτή η δυνατότητα θα μπορούσε να μειώσει το ποσοστό χρηματοδότησης από τον εθνικό προϋπολογισμό κατά ένα δις. Είναι σημαντικό ποσό. Και αντίστοιχη αύξηση της ε, κοινοτική χρηματοδότησης. Η πρότασή μας που είναι σε συντονισμό και με τις προτάσεις για το γενικό κανονισμό για τα διευθυντικά ταμεία αλλά έχει λοιπόν συμφωνηθεί να υπάρξει και την επόμενη περίοδο προγραμματισμού αυτό το topping up για να υπάρχει μια συνέχεια. Δεν θα υπάρχει λοιπόν καταληκτική ημερομηνία όπως υπάρχει τώρα για να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση στη νέα κατάσταση του νέου κοινού κανονισμού τρόπου εφαρμογής. Επέκταση λοιπόν του topping up μέχρι τέλος της περίοδου προγραμματισμού. Αυτά είχα να πω γι' αυτό. Το δεύτερο Το δεύτερο λοιπόν είναι ο κανόνας για την ε, αποδέσμευση. Σχετίζεται και αυτό με τις πολιετές ε, δημοσιονομικές προοπτικές, γιατί υπάρχουν κάποιες προβλέψεις εκεί Όταν μιλάμε για την χορήγηση πιστώσεων προς τα κράτη-μέλη, υπάρχει το λεγόμενο αντίστροφο δίκτυο ασφαλείας. Δηλαδή την επόμενη περίοδο τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να λάβουν περισσότερο από 110% των ε, πιστώσεων που, θα έχουν λάβει κατά την τρέχουσα. Οι διατάξεις αυτές ε, έχουν επιπτώσεις για δύο κράτη-μέλη, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. τι έλεγε το σχέδιο πολιτών προοπτικών του Φεβρουαρίου. Η Κομισιόν είχε προσκληθεί να διερευνήσει πρακτικές λύσεις για αυτές τις δύο χώρες, ούτω ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος αποδέσμευσης και να τροποποιηθεί ο παρόν κανονισμός των διαθροτικών ταμείων 1083. Συνεργαστήκαμε με τα δύο κράτη-μέλη πολύ στενά εξετάσαμε μια σειρά από λειτουργικές και τεχνικές λύσεις, επιχειρησιακές και τεχνικές λύσεις, για να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος αποδέσμευσης και διαπιστώσαμε ότι δεν θα μπορέσουμε να μειώσουμε αυτό το κίνδυνο κάτω από ε, ένα συγκεκριμένο επίπεδο που είναι αρκετά υψηλό για τη Ρουμανία. Προτείνουμε λοιπόν τροποποίηση του κανονισμού του Γενικού Κανονισμού Διαθροτικών Ταμείων του Ισχύοντος. Κατά την εξέταση του θέματος αυτού θεωρήσαμε ότι ο απλούστερος τρόπος θα είναι να επεκταθεί το 1 συν 3 ε, στις ε, πιστώσεις υποχρεώσεων του 11, 12 κτλ. Έτσι λοιπόν καταργούμε τους διπλούς στόχους ε, υποχρεώσεων για φέτος. Έτσι λοιπόν και του 12 θα πάει στο 15. Και έτσι θα βοηθήσουμε τις δύο αυτές χώρες, θα τους, δίσουμε, θα τους δώσουμε περισσότερο χρόνο να ε, υλοποιήσουν προγράμματα Στόχος μας είναι πάντα να είναι εφικτά αυτά που αποφασίζουμε, να μπορέσουν να εφαρμοστούν από τα κράτη-μέλη και είμαστε πεισμένοι ότι η πρόταση αυτή θα μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο αποδέσμευσης. Τώρα το τελευταίο σημείο είναι αν έχουμε χρόνο. Ξέρω ότι το μεγαλύτερο, το ευρύτερο νομοθετικό πακέτο είναι σε συζήτηση μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και θέλω να τονίσω ότι αναφερόμαστε και στο μέλλον τον κανονισμό της επόμενης γενιάς τον κοινό κανονισμό, τον κοινό εφαρμοστικό κανονισμό για όλα τα ταμεία θεωρούμε ότι πρώτα θα πρέπει να εγκριθεί ο γενικός κανονισμός και μετά ή επιμέρους, αλλά όλα αυτά πριν από το τέλος του χρόνου. Θα πρέπει να γίνουν ε, αλλεπάλια αυτές ε, οι εγκρίσεις, ε, αλλά πριν το τέλος του χρόνου. Γιατί υπάρχει ένα θέμα στο γενικό κανονισμό σε σχέση με την κατάργηση του 1083, άρα θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν από το φθινόπωρο μέχρι τέλος του έτους. Νομίζω ότι είναι σκόπιμο να το αναφέρω και αυτό. Και οποιασδήποτε τεχνικές λεπτομέρειες με χαρά να τις εξετάσω. Πρόεδρος. Το Φεβρουάριο υπήρξαν κάποιες αποφάσεις, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς ε, τι ακριβώς θα αποφασίσουμε για το γενικό κανονισμό, γιατί αυτό το τμήμα δεν το έχουμε αποφασίσει ακόμα, είναι πολιτική απόφαση. Ο Ότσιχ. Λοιπόν, θα μιλήσω τσεχικά. Θέλω πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω το σημευτό της της ημερήσιας διάταξης. Επειδή αύριο θα γίνει μια διάσκεψη για την πολιτική συνοχή στην Πράγα και θα συμμετέχω. Δεν μπορούσα να είμαι αύριο, οπότε και προβλεπόταν το θέμα. μου. Θα συζητηθεί λοιπόν σήμερα και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ακούσαμε λοιπόν ε, στην παρουσίαση του εκπροσώπου της Επιτροπής συγκεκριμένα στοιχεία. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Τα διαρθρωτικά ταμεία έχουν ε, δημιουργηθεί κατά τρόπον ώστε να παρέχουν βοήθεια στα μεμονωμένα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να εξέλθουν από την κακή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Και βέβαια κυρίως να εξέλθουν από την κρίση και να δημιουργηθούν εκ νέου χωρίς αυτές οι συνθήκες για ανάπτυξη. γίνονται βήματα προς την κατεύθυνση μετασχηματισμού. Ρουμανία και Βουλγαρία είναι οι χώρε, Ιταλία, Μάλτα, Τσεχία, Δανία, Σλοβακία που έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα και άλλε. Ε, αυτά τα βλέπετε σε ένα πίνακα Επομένως δεν μιλάμε μόνο για τις δύο χώρες που προαναφέρθηκαν. Αν θέλουμε λοιπόν να βρούμε την κατάλληλη λύση στο πρόβλημα, το πρώτο σκέλος του μέτρου, δηλαδή το top-up, αυτή η συμπληρωματική χρηματοδότηση θα ήταν μια καλή λύση. Δηλαδή, ε, μείωση κατά 10% του ποσοστού συγχρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη, όταν δεν υπάρχουν ε, δηλαδή κονδύλια για τη συγχρηματοδότηση ορισμένων ε, έργων και σχεδίων στον προπολογισμό των κρατών μελών. Δεν έχω λοιπόν κάποια αντίρρηση. Δεν θέλω να αναφερθώ μεμονωμένα ε, σε κράτη-μέλη. Αναφέρθηκαν διάφορες χώρες προηγουμένως. Το μέτρο αυτό πάντως έχει αποδειχθεί ότι είναι κατάλληλο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει τώρα να το επεκτείνει και στην, και στην επόμενη περίοδο ώστε να υπάρχει μια συνέχεια. Και όποιο κράτος μέλος ε, μπει σε συνθήκες μνημονίου θα μπορεί να αποφεληθεί από αυτό το αυξημένο, από την πλευρά την κοινωτική δηλαδή, ποσοστό συγχρηματοδότησης πάντοτε ε, το ζητούσαμε από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζητούσαμε και κάποιες εξαιρέσεις, οπότε τώρα θα έλθω στο δεύτερο σκέλος ε, του μέτρου, που είναι ο κανόνας νησιν 2 νησιν 3. Νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς συστημικό το ότι για τα πρώτα χρόνια όλα τα κράτη μέλη υπόκεινται στον κανόνα νησιν 3. Για τα έτη 2011-2012 όμως στον κανόνα νησιν 2. Η Σλοβακία και η Ρουμανία έχουν εξαίρεση, μπορούν δηλαδή να χρησιμοποιήσουν το κανόνα νησιν 3 για την όλη αυτή περίοδο. Προσωπικά πιστεύω ότι όχι μόνο όταν λόγω δύο κράτη-μέλη αλλά και άλλα κράτη θα έπρεπε να έχουν χρόνο ώστε να μπορέσουν να επιλέξουν τα βέλτιστα προγράμματα, σχέδια. Οπότε η ταυτόχρονη χρήση των δύο κανόνων, νήσιν 2, νήσιν 3 για τα έτη 2013-2014 θα δυσκόλευε την εξέβριση, την άλυση χρηματοδότηση από αυτά τα κράτη. Ένα άλλο σημείο που θέλω να αναφέρω Σε ό,τι αφορά το πολιτές μεσονομικό πλαίσιο, ακόμη οι εξελίξεις δεν είναι σαφείς, υπάρχει ρευστότητα και ενδεχομένως θα υπάρξει καθυστέρηση. Η επέκταση λοιπόν του κανόνα από νη 2 σε νη 3 για όλα τα κράτη-μέλη πιστεύω ότι θα μας βοηθούσε να μην έχουμε πρόβλημα στο πρώτο κομμάτι της περίοδου 2014-2020. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα σε ορισμένα κράτη-μέλη, ορισμένα έχουν ε, υποστεί πολύ μεγάλες πλημμύρες, οπότε η, χρήση του κανόνα που ίσχυσε για το 2011 και 2012 θα μπορούσε Το νησιν 3 δηλαδή να ισχύσει και σε αυτή την περίπτωση, να επεκταθεί χρονικά. Αυτή την περίοδο νησιν 3 Κομισιόν σκοπεύει να τη χρησιμοποιήσει για όλα τα κράτη-μέλη για την περίοδο 2014-2020. Γιατί να μην γίνει ήδη από τώρα, δηλαδή και για το 2011 και για το 2012. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Πιστεύω ότι με τη δική σας ε, συμβολή θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε μια λύση η οποία θα είναι αποφελής προς όλα τα κράτη-μέλη. Άρα όλα τα κράτη-μέλη θα μπορούν να αντλούν την χρηματοδότηση, τα κονδύλια. Δεν πρόκειται περί αύξησης της χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμο στα προγράμματα, αλλά μιλάμε ουσιαστικά για πλήρη αξιοποίηση των κονδύλων χρήση όλων των διαθέσιμων κονδυλίων. Πρόεδρος, δεν έχω ονόματα για τους σκιώδεις συγκητές, δεν ξέρω ποιοι είναι. Αν έχουν οριστεί σκιώδεις συγκητές από τις διάφορες πολιτικές ομάδες, να με ενημερώσετε η σοσιαλιστική ομάδα ποιον έχει ο σκιώδη, το Βίκτορ, το Βίκτορ Κωστινάρο, μάλιστα. Παρακαλώ, Βίκτορ. Madam Chair, if EPP... με μήπως θα έπρεπε να μιλήσει πρώτος ο εκπρόσωπος του ΕΛΚ. Μήπως δεν έχετε ορίσει σκιώδη γιατί... θα έρθει ο κύριος Ντόιτς, αλλά υπήρξε η αλλαγή στην ημερησία διάταξη και πώς μπορούν οι συνάδελφοί μου να γνωρίζουν ότι το θέμα Βλάσακ θα έρθει πρώτον. Αυτό ήταν μια έκπληξη για μας. Έχω σοβαρές αμφιβολίες για το αν το θέμα αυτό παρουσιάζεται σαν μια τεχνική απλά ρύθμιση και αν σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να διευρύνουμε την εμβέλειά του κατά τη διάρκεια της νέας περίοδου. Το θέμα φαίνεται πρακτικό, τεχνικό, αλλά από ό,τι κατάλαβα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το θέμα είναι να βρούμε μία λύση έτσι ώστε τα ταμεία να δουλέψουν πραγματικά όπως θα έπρεπε. Δεν ξέρω ποιες είναι, εν πάση περιπτώσει, οι προθέσεις μας, αλλά δεν ξέρω αν και η μέθοδος που ακολουθούμε είναι η σωστή. Και δεν θα πρέπει να θεωρήσετε ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα συμφωνήσει ακόμα και αν δεν εκφραστεί. Κοιτάξτε, για την ενημέρωση της ημερήσιας διάταξης ενημερώθηκαν όλοι οι σκιώδεις εισηγητές και οι συντονιστές από τη γραμματεία. Ο κύριος Μποστινάρου έχει το λόγο. Λίγες παρατηρήσεις. Πρώτον, ναι. Είναι προφανές ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καλή, έρχεται έγκαιρα και μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα πριν είναι πια αργά. Δεύτερον, είναι γεγονός πλέον ότι οι δύο χώρες οι οποίες θίγονται περισσότερο από την κρίση αντιμετωπίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτόν τον τρόπο και αυτό ήταν κάτι που βοήθησε ιδιαίτερα για τις ε, χώρες αυτές και τις περιφέρειές τους. Και τρίτον, οι δύο χώρες όπου οι μόνες οι οποίες επηρεάζονται από το διπλό κάπινγκ, πρέπει να το ξαναπούμε αυτό, πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας πριν περάσουμε σε οποιαδήποτε άλλη αξιολόγηση της απόφασης του Συμβουλίου, πριν συζητήσουμε άλλα θέματα, και να δούμε γιατί μόνο η Ρουμανία και η Σλοβακία συνέβη αυτό και όχι και σε άλλες χώρες. Τέλος, η απόφαση που πήρε εκείνη τη νύχτα, τη μεγάλη νύχτα, το Συμβούλιο, η απόφαση ελήφθη ομόφωνα. Ομόφωνα. Όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ήσαν παρόντες. Ο αρχηγός της Ρουμανίας δεν ήταν παρόν στη συγκεκριμένη συζήτηση, αλλά αυτή είναι η απόφαση στην οποία κατέληξε επίσημα το Συμβούλιο και γι' αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και να το σεβαστούμε. Τέταρτον, υπάρχουν κάποιες, κάποια θέματα, πραγματικά ουσιαστικά ειλικρινή θέματα, γιατί μόνο να είναι δύο οι χώρες αυτές, Σλοβακία και Ρουμανία. Εξ ονόματος της ομάδας θα ήθελα να πω ότι η αναθεώρηση η οποία προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σαφώς συνακτική με την απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο και επιτρέπει στις δύο συγκεκριμένες χώρες να επηρεαστούν λιγότερο από τις αποδεσμεύσεις. Από ό,τι φαίνεται η Ρουμανία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής θίγεται περισσότερο από τις αυτόματες αυτές αποδεσμεύσεις. Οι απώλειες είναι τεράστιες και είναι ελάχιστες οι δυνατότητες ανάκτησης εάν δεν περάσει το συγκεκριμένο μέτρο. Και η δεύτερη χώρα η οποία φύγεται είναι η Σλοβακία. Και τέλος να μου επιτρέψετε να αναφέρω και κάτι περισσότερο. Στην προπαρασκευαστική φάση για την τροπολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγιναν συζητήσεις και σε επίπεδο κορεπέρ. Οι συζητήσεις αυτές είχαν σαν στόχο την διεύρυνση του αριθμού των κρατών μελών που μπορούν να επωφεληθούν από την ρύθμιση. Στην αρχή μιλάγαμε μόνο για Σλοβακία και Ρουμανία. Αυτές ήταν οι χώρες που συνεργάστηκαν με την Επιτροπή. Όμως η Επιτροπή εξέτασε τα θέματα αυτά, έλαβε υπόψη όλες τις αξιολογήσεις και εκτιμήσεις και χρηματοπιστωτικές και οικονομικές προσπάθησαν τα κράτη-μέλη και οι υπηρεσίες τους να προσπαθήσουν να δούνε τι επιπτώσεις θετικές ή αρνητικές θα υπήρχαν από την τροπολόγηση του κανονισμού και μετά από όλα αυτά θεωρώ ότι η μοναδική δυνατότητα την οποία έχουμε πλέον μπροστά μας είναι να εμείνουμε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να την υιοθετήσουμε το ταχύτερο δυνατόν έτσι ώστε να είναι εφαρμόσιμη άμεσα για τη Ρουμανία και την Σλοβακία και να αποτρέψουμε μελλοντικές αρνητικές επιπτώσεις στις διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του πολιετούς. Υποστηρίζω πλήρως λοιπόν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είμαι διατεθειμένος να συνεργαστώ και με τους υπόλοιπους συναδέλφους με τον εισηγητή έτσι ώστε σε έφετο χρόνο να καταλήξουμε στη σωστή απόφαση. Πριν ζητήσω τους φιλελευθέρους να πάρουν το λόγο, θα ήθελα να πω ότι καλό θα ήταν να μας ε, ε, πείτε γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο μέσο για να ε, εξυπηρετήσετε κατά κάποιο τρόπο την πολιτική απόφαση του Συμβουλίου. Τι ανάλυση κάνατε έτσι ώστε να καταλήξετε στη συγκεκριμένη πρόταση. Η κυρία Μανέσκου, εξ ονόματος των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ. Θα ομιλήσω την Ρωμανική. Βλέπω ότι έχουμε Ρουμανική διευμηνία. Όπως υπόθηκε και από τον συνάδελφο Μποστινάρο, είναι προφανές ότι η Ρουμανία και η Σλοβακία είναι δύο χώρες οι οποίες έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερως από την κρίση και από, από το διπλό κάπινγκ. Είναι επίσης αλήθεια ότι η Ρουμανία και η Σλοβακία είναι οι χώρες οι οποίες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει ορισμένες λύσεις έτσι ώστε να ξεπεραστεί το θέμα. Και ζήτησαν από την Επιτροπή να προσπαθήσει έτσι ώστε να αποτραπεί η αποδέσμευση για τα περιφερειακά ταμεία. Υποστηρίζω λοιπόν την πρόταση διεύρυνσης της ισχύω του κανονισμού, του κανόνα μάλλον μη συνδύο για τη Σλοβακία και τη Ρουμανία, κάτι το οποίο θα προσφέρει στις χώρες αυτές περισσότερο χρόνο, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν σωστά τα χρήματα της πιστώσης στα πλαίσια της εφαρμογής του προϋπολογισμού. Το συγκεκριμένο μέτρο το οποίο έγινε δεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιτρέπει περαιτέρω ευελιξία για τις δύο αυτές χώρες σε σχέση με τις δαπάνες που αποφασίζουν και σε σχέση με την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Ταμείων και δίνει τη δυνατότητα στις χώρες αυτές να έχουν περισσότερο χρόνο για την επιλογή των στρατηγικών προγραμμάτων τους. Γνωρίζω ότι τα περισσότερα από τα προγράμματα αυτά αναφέρονται σε θέματα ανταγωνισμού, ούτε κίνητρα για τις μικρομεσαίες και για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους νέους. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν το, επί, το είδος αυτών των προγραμμάτων που θέλουν να εφαρμόσουν οι δύο χώρες μέλη, βλέπουμε ότι έχει σημασία η λύση την οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνει δεκτή το ταχύτερο δυνατόν. εκτιμούμε το ότι το Συμβούλιο ομόφωνα υποστήριξε τη συγκεκριμένη πρόταση και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να χάνουμε πλέον χρόνο και να επανέλθουμε στη συζήτηση από την αρχή στο Συμβούλιο και να χάσουν έτσι την ευκαιρία οι δύο αυτές χώρες να λύσουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Θεωρώ ότι ο κύριος Βλάσακ υποστηρίζει την άποψη αυτή και πρέπει να πούμε ότι κάτι τέτοιο δεν επηρεάζει καθόλου τις πιστώσεις υποχρεώσεων. Δεν υπάρχει καμία πρόταση για την αλλαγή των μέγιστων πιστώσεων, των, του ανωτάτου ορίου και δεν υπάρχουν επιπτώσεις οικονομικές σε σχέση με τις πιστώσεις πληρωμών. Πρόκειται λοιπόν για μια πολιτική απόφαση η οποία θα λειτουργήσει θετικά στο επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών για τις δύο αυτές χώρες τα επόμενα χρόνια και όπως είπε και ο συνάδελφος Μποστινάρο, έχει σημασία τα μέτρα αυτά να υιοθετηθούν το ταχύτερο δυνατόν. Υποστηρίζω λοιπόν τον κύριο Βλάσσα και την πρότασή του. Ευχαριστώ Μπρεζίνα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά συμφωνώ με το ότι η Ρουμανία και η Σλοβακία είναι κράτη-μέλη που ζήτησαν αυτή την αλλαγή, ε, να περάσουν δηλαδή από τον κανόνα νη συν στον κανόνα νη συν Και νομίζω ότι αν δεν είχαν μεσολαβήσει αυτά που έγιναν μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου και τη σήμερα, ούτε κι εμείς ε, θα ε, μάλλον και εμείς θα είχαμε στηρίξει το, και ζητήσει το ίδιο μέτρο για την Τσεχία. Έχει γίνει πάντως το αίτημα της αλλαγής αυτής ε, από τις δύο χώρες ε, Ρουμανία και Σλοβακία. Υπήρξαν όμως πλημμύρες στην Τσεχία έκτοτε. Εμείς δεν θα είχαμε πρόβλημα στην Τσεχία με τη χρηματοδότηση. Θα μπορούσαμε να είχαμε παραμείνει στον κανόνα νησιν 2, αλλά προέκυψαν οι πλημμύρες. Επίσης, ε, οι χώρες, ε, οι πλέον πληγήσεις χώρες από τις πλημμύρες, πιστεύω ότι πλέον θα πρέπει να ε, μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν κονδύλια από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Και προσωπικά θεωρώ ότι όχι μόνο αυτά τα κονδύλια, αλλά και με άλλους τρόπους θα πρέπει να βοηθηθούν οι χώρες αυτές. συνάδελφοι από τη Ρουμανία και τη Σλοβακία ανησυχούν, ε, το κατανοώ αυτό, ότι ενδεχομένω αυτό περιπλέξει τα πράγματα και τι διαπραγματεύσει. αλλά παρακαλώ όλους να δείξετε κατανόηση, γιατί και εμείς δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την κατάσταση στην οποία σήμερα βρισκόμαστε. Ευχαριστώ.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 το συζητήσουμε τον Οκτώβριο και να το ε, αποφασίσουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά υπάρχουν δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι αυτό το ανώτατο όριο, το κάπινγκ για το μέλλον, για τη μελλοντική περίοδο, που θα μειωθεί για τη Ρουμανία και την ε, Σλοβακία. Γι' αυτό είναι τόσο περίπλοκη η κατάσταση. Γιατί σύμφωνα με την αρχική ε, διατύπωση, τα ποσά για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού είχαν υπολογιστεί υψηλότερα. Η Κομισιόν επίσης ανέφερε τον κίνδυνο αποδέσμευσης, μη χρήση δηλαδή κάποιων πόρων που έχουν ε, προγραμματιστεί για αυτές τις χώρες. Άρα το σημαντικό είναι τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο και η Επιτροπή ε, έκαναν κάποιες διαπραγματεύσεις και οι χώρες αυτές ε, εξέτασαν την κατάστασή τους μαζί με την Κομισιόν και υπήρξε και ε, συνένεση από πλευράς ε, Συμβουλίου και Επιτροπής για να πάρουν λοιπόν η Σλοβακία και η Ρουμανία αυτές τις περαιτέρω δυνατότητες να υποφεληθούν από την αλλαγή των ε, κανόνων ώστε να περάσουμε στο 1 3. Πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτό συνολικά δεν σημαίνει ότι θα αυξηθεί συνολικά το κονδύλι, απλώς θα μας επιτρέψει να εφαρμόσουμε προγράμματα υψηλής ποιότητας. Και αυτό που είναι επίσης πολύ σημαντικά, σημαντικό είναι ότι υπήρξε ομόφωνη ε, έγκριση αυτού του Συμβουλίου. Εάν ε, τώρα πρόκειται για θέμα ε, επέκταση και σε άλλες χώρες, αυτό πρέπει να μας το πει η Επιτροπή. Ο κύριος Χρυσόγελος. Ε, πράγματι η κρίση και οι πολιτικές που έχουν ακολουθεί έχουν δημιουργήσει αρκετά προβλήματα και στην απορρόφηση και στην υλοποίηση προγραμμάτων ε, και έχουμε και αρκετές καθυστερήσεις. Ένα βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν είναι εύκολο σε μια περίοδο κρίσης και ο δημόσιος τομέας αλλά και ο ιδιωτικός τομέας να βρει συγχρηματοδότηση. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και στους δημόσιους φορείς. Και το δεύτερο είναι ότι πολλές φορές δημιουργήθηκαν προβλήματα και καθυστέρησαν την υλοποίηση έργων. Επομένως, σε, γενικές σε γενική βάση είμαστε υπέρ της των αλλαγών αυτών που προτείνονται. Θα έλεγα όμως εν συντομία ότι πρέπει να έχουμε και υπόψη και δύο προβλήματα που είναι σοβαρά. Το γεγονός είναι βέβαια ότι θα ορισμένα προγράμματα επιφορηθούν με το 90% αλλά επειδή δεν αλλάζει ο συνολικός προϋπολογισμός αυτό σημαίνει ότι προγράμματα θα κοπούνε. Θα μειωθούν προγράμματα. Αλλά τα ίδια λεφτά με μεγαλύτερη συμμετοχή αρκετά προγράμματα κάποια προγράμματα θα ολοκληρωθούν, αλλά κάποια άλλα πρέπει να κοπούν εντελώ γιατί δεν βγαίνει ο προπολογισμό. Μειώνεται ο προπολογισμό. Και επίση ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι το νήσιν 3, δηλαδή ότι δίνεται παράταση τρία χρόνια αντί για δύο, σημαίνει ότι τα χρήματα θα έρθουν σε μεγαλύτερη διάρκεια. Δηλαδή θα έχουμε χρήματα ε, τα οποία θα κατανοηθούν σε τρία χρόνια αντί για δύο. Και αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα σε χώρες που είναι ήδη σε κρίση αναέτος θα είναι μικρότερο, μικρότερο ποσό που θα πάρουν τα κράτη-μέλη ε, γιατί θα είναι το νησιν 3 και δεν είναι το νησιν 2. Παρ' όλα αυτά θα είμαστε θετικοί στην ψήφιση των αλλαγών αυτών, απλώς επισημαίνω ότι υπάρχουν και αυτά τα σημαντικά προβλήματα. Ευχαριστώ. Thank you. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι δύσκολη κατάσταση και ιδιαίτερα ο και κάποιοι άλλοι. Δεν είμαστε από τον Άρη, είμαστε από συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Ορισμένα ενδιαφέρονται, ορισμένα κράτη-μέλη ενδιαφέρονται για να υπάρξει λύση. Ορισμένοι θέλουν να ενταχθούν σε αυτή τη λύση, άλλοι δεν ενδιαφέρονται. Οπότε εμείς ως Ρέτζι δεν θα αποφασίσουμε ποιος έχει δικαίωμα να λάβει συμπληρωματική συγχρηματοδότηση και ποιος όχι. Γι' αυτό η ερώτηση της Προέδρου μας προς την Επιτροπή είναι σκόπιμη. Ή θα υπάρχει ένας ε, αντικειμενικός κανόνας με τον οποίο επιλέγονται οι χώρες. Δεν είναι λοιπόν κατά τύχη οι δύο αυτές χώρες ε, στο, στη ρύθμιση αυτή ή εάν τελικά θα αποφασίσουμε να βάλουμε και άλλες χώρες. Για παράδειγμα, ε, λόγω πλημμυρών, όπως είπε ο συνάδελφος. διότι όπως καταλαβαίνετε αυτό θα επηρεάσει πολύ τις επόμενες πολιτικές προοπτικές. Συμπεριλήφθηκε στον συμβασμό γιατί έγινε ο υπολογισμό με βάση το δίκτυο ασφαλείας. Εάν έχουμε στοιχεία αντικειμενικά από την Κομισιόν, να υποστηρίξουμε τα στοιχεία, τη σωστή βάση. Δεν θα υποστηρίξουμε την ΑΒ χώρα. Θέλω λοιπόν να μας πει η Κομισιόν γιατί αυτές οι χώρες δεν είναι τυχαίο το ότι συμφώνησαν όλες οι χώρες συμφώνησαν με βάση κάποιους υπολογισμούς. Να μην αρχίσουμε τώρα να ε, φιλονικούμε για το ποιος του αξίζει. Κοιτάξτε, εγώ υπερασπίζομαι τις πολιτικές προοπτικές γιατί είναι καλές για την Πολωνία και εγώ είμαι Πολωνός. Αυτό μπορεί να ισχύει, αλλά δεν θα πρέπει να τσακωθούμε για, με τέτοια κριτήρια. Φρανσουά Αλφονσί. Η ομάδα μας υποστηρίζει αυτή την προσπάθεια. με εκπλήσει κάπως, με μπερδεύει κάπως η δυσχέρεια να εφαρμόσουμε ένα μέτρο που είναι προφανές, δεν είναι. Και που ε, αφισβητεί και την ε, μακροοικονομική ερεσιμότητα. Υπήρξαν πλημμύρες. Αλλά δεν αντιμετωπίζουμε συγκυριακά προβλήματα, αντιμετωπίζουμε πιο ουσιώδη προβλήματα, οικονομική κρίση και πώς θίγει ορισμένες χώρες και διαπιστώνουμε ότι η μακροοικονομική αιρεσιμότητα λειτουργεί αντίστροφα. Και είναι λογικό. Αντί να λειτουργεί όπως μας την πρότειναν, ως κύρωση για τις χώρες που έχουν μεγάλες δυσχέρειες, διαπιστώνουμε ότι όσο μεγαλύτερες δυσχέρειες έχει μια χώρα, τόσο περισσότερο πρέπει να τη βοηθήσουμε να απορροφήσει τους πόρου με πιο ελαστικού, πιο προσαρμοσμένου κανόνε. Πιστεύω λοιπόν και συμμερίζομαι τον ε, τελευταίο ομιλητή, οι αποφάσεις μας δεν πρέπει να είναι συγκυριακές. Πρέπει να είμαστε συστηματικοί. Όταν υπάρχουν τέτοιου τύπου δυσχέρες να λέμε, όταν αποδεικνύεται ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη να αξιοποιηθούν περισσότερο οι ε, ευρωπαϊκοί πόροι, ε, να γίνεται με μεθοδικό τρόπο, όχι τυχαία και ανάλογα με την καλή θέληση της τάδε συνάντησης του Συμβουλίου, που συζητάει τόσα και τόσα θέματα στην ημερήσια διάταξη του κάθε φορά. Πρόεδρος. Γιώχη Μτσέλα. Ευχαριστώ. Προχθές πήραμε πάλι μια επισκόπηση για το ποσοστό πληρωμών για κάθε χώρα και είναι πολύ διαφοροποιημένη η εικόνα για το ποιες πληρωμές, πόση απορρόφηση, ποιες υποχρεώσεις και πάντα οι ίδιες χώρες είναι στις τελευταίες θέσεις. Εξάλλου, από τότε που είμαι ευρωβουλευτής, πάντα τίθεται το ερώτημα ε, εάν και κατά πόσο πρέπει να υπάρξουν διευκολύνσεις και ελαφρύνσεις για κάποια κράτη, συμπληρωματικές συμφωνίες, νέοι κανόνες, για να μπορέσουν να απορροφήσουν καλύτερα τα κονδύλια που είναι στη διάθεσή τους. Το 2010, θυμάστε, συζητήσαμε και αποφασίσαμε ότι για ορισμένα κράτη-μέλη οι ενισχύσεις από το δικό τους προπολογισμό, το ποσοστό δηλαδή συγχρηματοδότησης, μπορεί να επιστρέφεται ή να μειούται. Τότε, πέρσι, με πρωτοβουλία της Προέδρου μας, δημιουργήσαμε αυτό το μέσο ε, Κατανομή των κινδύνων για να μπορούμε να χρηματοδοτούμε μακροπρόθεσμα προγράμματα και να υπάρχει δυνατότητα ακόμη και πλήρους χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους. Όταν ε, πτωχεύουν κάποια ιδρύματα που είχαν ε, ή κάποιοι ιδιωτικοί χρηματοδότες που είχαν ε, υποσχεθεί ε, να συμμετάσχουν. Τώρα θέλουμε να βοηθήσουμε κάποια κράτη να αξιοποιήσουν καλύτερα κάποιες χρηματοδοτήσεις επειδή είδα την κατάσταση στα συγκεκριμένα αυτά κράτη, έχω την υποψία ότι δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων, να υπάρχουν δηλαδή διαθέσιμες πιστώσεις, ότι, αλλά ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν προβλήματα ε, διαχείρισης των προγραμμάτων. Δεν υπάρχουν οι διοικητικές δομές, δεν έχουν αναπτυχθεί, ούτως ώστε να εφαρμόζονται με συνέπεια προγράμματα και τα, ε, οι πιστώσεις να αξιοποιούνται σωστά και αποτελεσματικά Παίζουν ρόλο και αλλαγέ κυβερνήσεων, διότι ε, οι κυβερνήσει αποφασίζουν ποια προγράμματα θα χρηματοδοτούν και ποια όχι και μετά οι κυβερνήσει και τα προγράμματα. Νομίζω λοιπόν ε, ότι δεν είμαι σίγουρο ότι είναι καλέ προτάσει αυτέ τη Επιτροπή. Πρόεδρο. Ήβα Κούντμαρς Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για αυτό το θέμα είναι σαφέστατο ότι η σύνοση πρέπει να βοηθήσει αυτούς που έχουν θυγεί περισσότερο. Το γράφει η συνθήκη. Τι σημαίνει συνοχή. Προσπαθείς αυτός που είναι πιο αδύναμος να, να πλησιάσει τους ισχυρότερους. Αυτό το δήμα του διπλού ανώτατου ορίου double capping θα το αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον. Γιατί είναι σαφές. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι μεγάλες χώρες που έχουν πολλές περιφέρειες με διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης. Και το ΑΕΠ ε, δεν είναι λιγότερο από το 75% ή μεταξύ 75 και 90 μετάβασης θα εφαρμόσουν αυτόν τον τύπο αλλά τελικά θα υπάρξει το όριο λόγω του ε, συνολικού ΑΕΠ της χώρας. Ενώ οι μικρότερες χώρες που έχουν μόνο μία περιφέρεια δεν έχουν καμία τέτοια δυνατότητα. Είναι πρόβλημα αυτό το ανώτατο όριο, αλλά τι άλλη λύση να βρούμε. Γιατί βασίζεται στο ΑΕΠ. Η κατάσταση τώρα είναι διαφορετική από το 10 και Τότε αποφασίσαμε να βοηθήσουμε πέντε χώρες με 770 εκατομμύρια, ούτως ώστε να γίνουν ταχύτερα κάποιες ενδιάμεσες πληρωμές, κάποιες προκαταβολές αυτές τις χώρες οι πέντε χώρες ήταν εκείνες οι οποίες ελάμβαναν βοήθεια από το ΔΝΤ ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λέω μιλητής. Ε, τώρα εδώ δεν προτείνεται να δοθούν συμπληρωματικές πιστώσεις, αλλά να μπορέσουν να γίνουν σεβαστές οι υποχρεώσεις. Και υπάρχει ένα θέμα αρχής. Εγώ υποστηρίζω αυτή την πρόταση, γιατί βλέπω τη δυναμική της απορρόφησης από το 2007 κάθε μήνα και προσπαθώ να καταλάβω γιατί είναι τόσο διαφορετικός ο, τόσο διαφορετικό το ποσοστό απορρόφησης. Μίλησα και με την αντίστοιχη υπηρεσία της Κομισιόν και μου είπαν ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα ελέγχων, υπάρχουν προβλήματα ε, ποιότητας των προγραμμάτων και η Κομισιόν είναι πολύ αυστηρή. Δεν επιτρέπουν να προχωρήσει ένα πρόγραμμα πριν λυθούν αυτά τα προβλήματα. Σε πολλές χώρες. Καθυστερούν οι πληρωμές 6 ε, μήνες, 10 ε, μήνες, πάνω από χρόνο. Γι' αυτό το λόγο. Εάν αυτό το μέτρο θα επιτρέψει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες δομές χωρίς να αυξηθούν οι χρηματοδοτήσεις, το υποστηρίζω. Κοιτάξτε, αν πάτε στην Επιτροπή Προπολογισμών Κοιτάξτε βέβαια και στο νέο μας ε, κανονισμό υπάρχει το NC2 και το NC3. Δεν το αλλάζουμε. Αν έχουμε το NC3 για αυτούς που είναι λιγότερο ε, από 82% με βάση τον υπάρχοντα κανονισμό ή για κάποιες περιφέρειες νη συν 2 και δεν το έχουμε αλλάξει τον επόμενο κανονισμό ναι ναι εν συν 3 γίνεται άρα προσθέτουμε κάτι αλλά αν από τη μία δίνουμε με το ένα χέρι εν συν 3 ξέρουμε ότι τα προγράμματα είναι σοβαρά και δεν μπορεί να τελειώσει ένα πρόγραμμα συνοχής μέσα σε 7 χρόνια Άρα πρέπει να βρούμε κάποια λύση με τους υπεύθυνους του προπολογισμού. Δεν υπάρχει αυτή η διαφωνία επειδή δεν θέλουμε να υπάρξει απορρόφηση. Είναι η κατάσταση διαφορετική από χώρα σε χώρα. Ε, από τη Γερμανία, στη Λετωνία. Υπάρχουν κάποιες χώρες που έχουν καλύτερη απορρόφηση. Αλλά αυτό είναι αναπόφευκτο γιατί δεν είμαστε μια χώρα, είμαστε η Ευρώπη. Και ε, λόγω και της κρίσης τότε ε, υπάρχουν ακόμη ευρύτερες διαφοροποίησεις διότι οι επιπτώσεις της κρίσης είναι άνισες. Στη χώρα μου είχαμε μείον 24% σε δύο χρόνια. Ενώ σε άλλες ε, χώρες δεν έχει μειωθεί το ΑΕΠ. Λοιπόν, Μαθηματικά θα ήταν πολύ καλό να πούμε για όλες τις χώρες ο ίδιος κανόνας. Θα υπάρχει ο ίδιος χρόνος και αν δεν, αν δεν το επιτύχετε θα αφαιρεθούν οι χρηματοδοτήσεις. Αλλά η ζωή είναι διαφορετική, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Πρέπει να στηρίξουμε αυτό το μέτρο. Γιατί οι χώρες που θα αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα δεν θα πάρουν περισσότερες πιστώσεις, θα πάρουν περισσότερο χρόνο. Το θέμα είναι πώς θα το εφαρμόσει η Κομισιόν. δεν είναι δυνατόν η Κομισιόν ε, να έχει λειτουργήσει τόσο άσχημα. Και σας κατηγορώ συγκεκριμένα. Είναι πολύ περίπλοκο γιατί σταματάνε οι πληρωμές. Τέσσερα χρόνια εδώ μέσα δεν μας έχετε πει εσείς κύριε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε τις χώρες. Δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε και να καταδώσουμε κανέναν. Αλλά οι λόγοι μία απορρόφησης δεν έχουν αναλυθεί. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε ως ευρωβουλευτές. Δεν έχουμε τη σωστή πληροφόρηση. Εσείς την έχετε. Θα ήμουν ιδιαίτερα ευγνώμων εάν στο τέλος της περίοδου πολιετών προοπτικών μας δώσετε πληροφόρηση που να μπορέσουμε να δώσουμε στην επόμενη θητεία. Κορνέλια Έρνστ. Λοιπόν, οι δύο προτάσεις ε, που μας έγινε από την Επιτροπή πρέπει να τύχουν πλήρους υποστήριξης. Δεν είναι θέμα ποσοστών. Δεν θέλουμε να κάνουμε παζάρια. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Δεν χρειάζομαι ε, εξηγήσει γιατί οι χώρε αυτέ, οι προηγούμενε χώρε, η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, γιατί χρειάζονται topping up, το καταλαβαίνω. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αυτά που γίνονται στο Συμβούλιο με αυτά που κάνουμε εμείς. Μπορεί να κάνει λάθος το Συμβούλιο, που εμείς δεν μπορούμε να τα διορθώσουμε, αλλά πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δημιουργήσουμε περισσότερε δυνατότητε απορρόφησης. Και αν ε, ανακάμψουν αυτές οι χώρες, θα έχουμε κάνει κάτι σωστό. Είναι λογικό αυτό. Νομίζω ότι είναι απλώς θέμα συνέπειας το σημείο 2. Ήρθαν εδώ ε, ήρθε εδώ ο Πρωθυπουργό της Ρουμανίας και μας είπε ότι είναι αναγκαίο να γίνουν ε, μεταρρυθμίσεις στις δομές, ότι έχουν ξεκινήσει. Καταλαβαίνω τι σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε αλλαγές και εμείς στη Γερμανία κάνουμε πολλές αλλαγές, πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Και δεν είναι μόνο θέμα πλημμυρών σε κάποιες χώρες. Πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθεί η διακυβέρνηση, η διαχείριση των προγραμμάτων και πολλά άλλα. Γιατί όμως ε, πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η αλλαγή μόνο για τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Νομίζω ότι και σε άλλες χώρες ε, υπάρχουν παρόμοιες συνθήκες. Θα ήταν σκόπιμο να δοθεί περισσότερος χρόνος για να μπορέσουν να εφαρμοστούν τα πρόγραμμα. Πρέπει να υποστηριχθεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα διαφορετικό. Δεν έχω άλλους ομιλητές που να θέλουν το λόγο πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και θα ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάρα πολύ σύντομα να μας επαναλάβει γιατί οι δύο αυτές χώρες επελέγησαν στα πλαίσια της πολιτικής απόφασης του Συμβουλίου. Και θα ήθελα να μάθω πριν περάσουμε στις αλλαγές του κανονισμού, σκεφτήκατε και άλλου τύπου μέτρα, άλλου είδους μέτρα τα οποία θα βελτίωναν την απορροφητικότητα και θα μείωναν τις πιθανότητες αποδέσμευσης. Ευχαριστώ. Επανέρχομαι στο πρώτο σας αίτημα. Είναι κάτι το οποίο τέθηκε όμως στα πλαίσια των κριτηρίων τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν στα πλαίσια της συγκεκριμένη πρότασης. Καταρχάς συνειδητοποιούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η απορρόφηση. Αλλά προσπαθήσαμε να δούμε και κάποια σκεπτικά τα οποία θα έλεγα εξηγούν αν θέλετε την επιλογή της συγκεκριμένης παραγράφου. Οι δύο αυτές χώρες λοιπόν επηρεάζονται από ε, ένα ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό. Criteria and you will see that in recital uh, number 6 we make the reference to the Γίνεται μια αναφορά λοιπόν στις συγκεκριμένες αυτές χώρες. Τα κριτήρια ε, τα οποία χρησιμοποιήσαμε λοιπόν για την πρότασή μας είναι γνωστά. Αναλύσαμε ταυτόχρονα και τις διαφορετικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν για να μειωθούν και να αποτραπούν οι κίνδυνοι της αποδέσμευσης και για τις δύο αυτές χώρες αλλά και για άλλες χώρες. Θα ήθελα τώρα να επιμείνω λίγο περισσότερο στη δική μας αιτιολόγηση. Η λογική μας εδράζεται θα έλεγα στο, στις πολιετής προοπτικές και στις προβλέψεις μας για τις πολιετής προοπτικές σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι διαφορετικές επιλογές οι οποίες ε, μελετήθηκαν σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη αυτά, τα δύο κράτη-μέλη, αλλά και σε συνεργασία με εκπροσώπους άλλων κρατών μελών. Το πιο ε, θα έλεγα προφανές από τα θέματα πέραν του topping up είναι τα λεγόμενα ποσοστά συγχρηματοδότησης και ορισμένα λειτουργικά προγράμματα δεν βρίσκονται στο επίπεδο στο οποίο προεβλέπετο. Μελετήσαμε λοιπόν την δυνατότητα να αυξήσουμε τα ανώτατα νομικά όρια τα οποία προβλέπονται από το παράρτημα του Γενικού Κανονισμού. Ε, ένα αντισταθμιστικό ποσοστό δηλαδή. Άλλες επιλογές που κοιτάξαμε ήταν ο αναπρογραμματισμός ή εκ νέου προγραμματισμός. Πάρα πολλές φορές συμβαίνει κάτι τέτοιο και εδώ να υπογραμμίσω ότι τα τελευταία χρόνια προχωρήσαμε στη χρήση του μέσου αυτού έτσι ώστε να συλλέξουμε επενδύσεις σε κομβικούς τομείς, σημαντικούς τομείς για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, όπως επίσης και την δημιουργία καλύτερων ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης. Έχουμε ας πούμε και διάφορες πρωτοβουλίες στα πλαίσια των οποίων προχωρήσαμε σε εκ νέου προγραμματισμούς και στη Σλοβακία είναι μια επιλογή για τη μεταφορά πιστώσεων ανάμεσα σε προγράμματα και συνεργασία ανάμεσα σε προγράμματα. Εμείς δεν θέλουμε να καταστήσουμε ευκολότερη την συγχρηματοδότηση, αλλά θέλουμε να βοηθήσουμε τα προγράμματα έτσι ώστε να επιταχύνουν την οικονομική ανάπτυξη. Τώρα τα λεγόμενα μείζωνα προγράμματα. Βλέπετε ε, ε, ότι τα προγράμματα αυτά πράγματι θα πρέπει να είναι σωστά προπαρασκευασμένα. Εμείς τα προωθούμε με τον ταχύτερο τρόπο, συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη για τις δυνατότητες επιτάχυνσης ε, των ε, ε, ετοιμάτων για χρηματοδότηση προγραμμάτων μεγάλου μεγέθους. Και φυσικά αυτό δεν θα πρέπει να ξεπερνά και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον κανονισμό. Αυτό αφορά και άλλα θέματα. Βλέπουμε ας πούμε ότι τίθεται το θέμα της διοικητικής ικανότητας. Έχουμε αναπτύξει ορισμένα προγράμματα δράσης στα διάφορα κράτη-μέλη, στη Ρωμανία και στη Σλοβακία δηλαδή, έτσι ώστε να πετύχουμε πολύ συγκεκριμένους στόχους γύρω από δράσεις οι οποίες θα πρέπει να αναλυθούν για να επιτρέψουν τη σωστή ε, χρήση των διαθέσιμων πιστώσεων βελτιώνοντας τις διοικητικές ικανότητες, τις διαχειριστικές ικανότητες για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. Να πω και κάτι για την Ελλάδα βέβαια. Εμείς και στα πλαίσια του Task Force προσπαθούμε να διευκολύνουμε την βελτίωση της διοικητικής διαχειριστικής ικανότητας των υπηρεσιών. Ξεκινήσαμε με την κρίση αυτή το 2008 και υποθέταμε ότι δεν θα συζητούσαμε τα ίδια πράγματα το 2013. Ε, ε, τα θέματα αυτά είναι θέματα τα οποία μας αφορούν ιδιαίτερα. Ε, συνεργαζόμαστε με τη δημόσια διοίκηση της χώρας αυτής και άλλων χωρών έτσι ώστε να μην ε, ε, δαπανώνται χρήματα αν δεν υπάρχει μια σωστή διοικητική διαχειριστική ικανότητα από πλευράς των αρμόδιων ε, για τη συγκεκριμένη δαπάνη υπηρεσιών. Είναι προφανές λοιπόν ότι θα πρέπει να επιτρέψουμε τα προγράμματα αυτά να αναπτυχθούν σωστά. Να αναφερθώ τώρα στις πλημμύρες. Νομίζω ότι οι πλημμύρες, όλοι γνωρίζετε, ήμουν στην Πρατισλάβα μέχρι χθε. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχα πάει στη Γερμανία και στην Πράγα. Οι κεντροευρωπαϊκές πραγματικά πλημμύρες είναι πολύ σοβαρές. Υπάρχουν μέσα, αναφερθήκατε και στο Ταμείο Αλληλεγγύης, Φυσικά ανησυχούμε σχετικά με τις ποσοστώσεις ε, προς το ταμείο αυτό που μπορεί να μειωθούν. Αλλά παρόλα αυτά συνεργαζόμαστε με τις εθνικές διοικήσεις των εμπλεκομένων χωρών και δίδουμε συστάσεις για να βελτιώσουν ε, σωστά και με τεκμηριωμένο τρόπο τα αιτήματά τους έτσι ώστε να αποζημιωθούν. Δεύτερον, υποστηρίζουμε επίσης την χρήση των διαφορετικών ταμείων και τα μέσα τα οποία προβλέπονται για την πρόληψη των πλημμυρών. Όπως είδαμε και χθε στην Πρατισλάβα υπάρχουν κάποια ελαφρού τύπου ευέλικτα φράγματα που χρηματοδοτήθηκαν από τα διαφορετικά ταμεία στις όχθες του Δούναβη στην Πρατασλάβα και ε, φύγει λιγότερο η πόλη από ό,τι αντίστοιχες περιοχές και πόλεις στην Γερμανία ή σε άλλες χώρες. Και τρίτον, εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τους εκπροσώπους των κρατών μελών έτσι ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στα πλαίσια της εφαρμογής προγραμμάτων που στοχεύουν στην αποτροπή ζημιών από τις πλημμύρες. Όλα αυτά είναι θεμητά προβλήματα, τίθενται με θεμητό τρόπο και ε, πραγματικά θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε και να περιορίσουμε και τον κίνδυνο αποδέσμευσης εδώ γιατί υπάρχει φυσικά μία force majeure. Εξετάσαμε πάρα πολλές επιλογές για να μειώσουμε τον κίνδυνο της αποδέσμευσης και νομίζω ότι όλα αυτά θα τα συμπεριλάβουμε στις αποφάσεις. Να ευχαριστήσω τον Διευθυντή από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής, γιατί σχετικά με τις πλημμύρες συνειδητοποιούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να βοηθήσει και συνειδητοποιούμε επίσης ότι κάποια προγράμματα λόγω των πλημμυρών μπορεί να καθυστερήσουν. Κλείνοντας να πω ότι όπως είπε και ο εισηγητής δεν θέλουμε εμείς να αμφισβητήσουμε ε, τα αιτήματα τα οποία έχει καταθέσει η Ρουμανία και η Σλοβακία και στο Συμβούλιο και ουδήποτε αλλού. Νομίζω ότι όπως και στο παρελθόν θα πρέπει να, να μην υπερασπιζόμεθα μόνο αυστήρα τα εθνικά μας συμφέροντα, ιδιαίτερα σε επίπεδο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, αλλά τις αρχές μας. Και η μοναδική μου αντίρρηση στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι θα πρέπει να σεβαστούμε πάρα πολύ απλά τις βασικές αρχές. Αν θέλουμε τώρα να μιλήσουμε για τις συμπληρωματικές πιστώσεις, τα top-ups ε, σε συγκεκριμένα ποσοστά και στα πλαίσια των συγχρηματοδοτήσεων. Αυτό είναι ένα μέσο το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία και θα θέλαμε να το χρησιμοποιήσουμε το θέμα της συμπληρωματικής χρηματοδότησης και στο μέλλον. Και αυτό θα πρέπει ε, να συνδυαστεί και με την εφαρμογή του κανόνα νη 3. Έχει ήδη αποδείξει το πόσο επιτυχές είναι σαν σύστημα Και το θέμα αρχής το οποίο τίθεται είναι ότι οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να υπάρχουν θα πρέπει να λαμβάνονται συνεχώς υπόψη κατά τη διάρκεια της περίοδου όχι για τις δύο συγκεκριμένες χώρες μέλη αλλά για όλες τις χώρες μέλη. Ένα επιπλέον σχόλιο για ένα μέσο το οποίο δεν χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά σύμφωνα με τις διαθέσιμες στατιστικές και αναφέρθηκε σε αυτό ο Διευθυντής. Είναι το θέμα του επαναπρογραμματισμού Τη μεταφορά δηλαδή πιστώσεων από προγράμματα όπου δεν χρησιμοποιούνται σε άλλα προγράμματα. Αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ και πάρα πολύ καλά. Η Ιρλανδία το έχει κάνει αυτό. 45% των πιστώσεων έχουν τύχει αναπρογραμματισμού. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο ε, καλύπτει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των διαθέσιμων πιστώσεων και από ό,τι ακούω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει αρκετά ευνοϊκά την συγκεκριμένη επιλογή. Τέλος λοιπόν, θα ήθελα να ακούσω και τις δικές σας απόψεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. Η έκθεση προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 10 Ιουλίου. Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών θα πρέπει να είναι η 17 Ιουλίου και η ψηφοφορία σχετικά με την εντολή που θα δώσουμε σαν Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα πρέπει να είναι 23η ή 24η Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ Οιτσικ. Πρόκειται για τη μέθοδο της συναπόφασης. Πρόκειται για μια συγκεκριμένη νομική πράξη. Στο Συμβούλιο έχουν προχωρήσει από ό,τι φαίνεται και η ταχύτητα έγκρισης αν θέλεις εξαρτάται κυρίως από τη δική μας προσπάθεια. Για όλους αυτούς τους λόγους θα πρέπει εμείς ε, να καλύψουμε τις ανάγκες των κρατών μελών το ταχύτερο δυνατόν. Να ακολουθήσουμε το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχεις προτείνει και να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του μηνός Οκτωβρίου. Το χρονοδιάγραμμα αυτό λοιπόν προϋποθέτει ότι θα έχουμε την πρόταση στην επόμενη συνάντησή μας, την 10η Ιουλίου, για να μπορέσουμε να την ψηφίσουμε σε επίπεδο Επιτροπής τον μήνα Σεπτέμβριο. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα λοιπόν όπως το προτείνει και ο εισήγητης. Λοιπόν κλείνω το συγκεκριμένο θέμα. Να περάσουμε τώρα στη συζήτηση των προτάσεων εκθέσεων για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων. Ξεκινάμε με το γενικό κανονισμό. Uh, Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να ξεκινήσω εγώ με την πρώτη ανταλλαγή απόψεων ε, για την ε, κατάσταση σε ό,τι αφορά τον ε, κοινό κανονισμό. Τις διατάξεις δηλαδή για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και την κατάσταση του κανονισμού 1083. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε διάφορα πράγματα. Είμαστε εν μέσω της ε, περίοδου κατά την οποία είναι δυνατή κατάθεση τροπολογιών και εμείς ως εισηγητές αλλά και σε πολύ καλή συνεργασία και συντονισμό με τους σκιώδεις είμαστε πάντοτε ανοιχτοί να σας δώσουμε οποιαδήποτε απαιτούμενη πληροφορία. Πολλοί συνάδελφοι μάλιστα ήδη ήλθαν σε εμά για να τους ενημερώσουμε και να τους εξηγήσουμε περισσότερο τα πράγματα. Είναι ακόμη ανοιχτή λοιπόν η διαδικασία. Σε προηγούμενες ε, συναντήσεις σας έχουμε ενημερώσει και τώρα υπάρχει και ένας κατάλογος ε, των χρηστών τροπολογιών. Ε, σας εξηγούμε πώς έχει κατάσταση, πού έχουμε επιτύχει συμφωνία, πού γίνονται ακόμα διαπραγματεύσεις και που ακόμη δεν είναι ξεκάθαρη η εντολή, τέλο πάντων δεν έχουμε πετύχει του στόχους μας. Ο βασικός μας στόχος είναι να προετοιμάσουμε σωστά την ψηφοφορία του Ιουλίου. Και βέβαια δεν θα πρέπει να επαναλάβω τώρα πράγματα τα οποία εξήγησα την προηγούμενη φορά. Θα είμαι σύντομος λοιπόν. Τις τελευταίες ημέρες η δική μας επιτροπή είχε οργανώσει δύο αποστολέ, δύο αντιπροσωπείε. Εγώ προσωπικά πήγα στη Βόρεια Σουηδία. Τι είδα και τι ένιωσα εκεί. Είδα να υπάρχει κάποια συμμετοχή των περιφερειών ε, στην ε, προετοιμασία των ε, συμφωνιών εταιρική σχέση. Όμως, ποιο είναι το κρίσιμο σημείο. Οι περιφέρειες, οι πόλεις πρέπει να συμμετάσχουν ακόμη περισσότερο στο στάδιο αυτό. Υπάρχουν ζητήματα για τα οποία έχουμε συμφωνήσει και αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει πρέπει να εφαρμοστούν στα διάφορα κράτη-μέλη και αυτό να γίνει μέσα στους επόμενους μήνες. Επομένως, είναι σημαντικό και στην Επιτροπή μας να σημειώσουμε πρόοδο, οι ομάδες διαπραγμάτευσης, ώστε το συντομότερο δυνατόν να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και έτσι να μπορέσουμε να ψηφίσουμε τον Ιούλιο, όπως προβλέπετε, στη διάρκεια της Συνόδου Συγκεκριμένα, τον Έχουμε και τον, τον Οκτώβριο την ε, ψηφοφορία στο Στρασβούργο. Έτσι θα μπορέσουν να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2014. Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο είμαστε πλέον σε τροχιά, ε, σταθεροί, Έχουμε συμφωνήσει για, στρατηγικά, για το στρατηγικό προγραμματισμό, την εδαφική συνεργασία, τον έλεγχο, την επιλεξιμότητα, την ενημέρωση. Αυτά τα θεματικά, ε, αυτές οι θεματικές ομάδες έχουν κλείσει σε τριμερείς διαλόγους, έχουμε συμφωνήσει και πολύ σύντομα, αύριο συγκεκριμένα, έχουμε έναν ακόμα τριμερή διάλογο. Ελπίζουμε να πετύχουμε συμφωνία για τέσσερις ακόμα θεματικές ομάδες. Ένα σημαντικό υποσυζήτηση σημείο είναι τα μερίδια του έκτου και του κοινωνικού ταμείου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει στην πράξη να εγγυηθεί αυτό το 25% που έχει ψηφιστεί για τους στόχους του κοινωνικού ταμείου όπως τους έχουμε διατυπώσει. Ακριβώς λόγω των αλλαγών με τους νέους κανονισμούς υπάρχει πλέον η δυνατότητα να έχουμε έναν σταθερό ε, προϋπολογισμό που θα είναι εγγυημένος, εξασφαλισμένος για το κοινωνικό ταμείο. Και θα μπορούμε επίσης να έχουμε και μία ε, προσέγγιση πολλαπλών κονδυλίων, πολλαπλής χρηματοδότησης. Ε, έχουμε συμφωνήσει επί της θεματικής συγκέντρωσης, όπως γνωρίζετε, και βέβαια σε κάποιες χώρες χρησιμοποιούμε και το ΕΤΠΑ το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, πάντα στα πλαίσια της εντολής μας. Ελπίζω να συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό τώρα. Για το μέλλον, τι έχει απομείνει, τι έχει ουσιαστικά απομείνει. Υπάρχει μια μείζον διαφωνία σε ό,τι αφορά το, το θεματικό επίδοσης, performance reserve. Τα θέματα θα πρέπει να δαπανηθούν αργότερα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία, θα γίνονται πολλά σε επίπεδο κρατών μελών. Και επειδή το είπα και πριν, ενδεχομένως να μην φτάσουμε καν ε, σε δαπάνη των ποσών αυτών για την επόμενη επταετία. Και μετά όταν έχουμε μια κρίση μπορεί μετά το... τα επόμενα χρόνια να χρειαστεί να διαπραγματευτούμε κάτι. Και σίγουρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε τους ε, οικονομικούς πόρους, ε, πόσοι είναι διαθέσιμοι και θα συνεχίσουμε τελο πάντων τον αγώνα μας πάνω σε αυτό. Το μέσο για, την, ε, για το Connecting Europe είναι ένα ακόμα προβληματικό, αν και όχι τόσο προβληματικό. Έχουμε εδώ σημειώσει κάποια πρόοδο. Ένα άλλο σημαντικό είναι η λεγόμενη macro-conditionality, μακροαιρεσιμότητα. Και στο, στις συζητήσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ελπίζουμε να έχουμε θετική έκβαση σύντομα. Έχουμε τώρα ε, τις διαπραγματεύσει στο ανώτατο επίπεδο. Ελπίζουμε να είναι θετική έκβαση, παραλαμβάνω. Στη δική μα Επίτροπη, ως συνομοθέτε, έχουμε και εμεί ευθύνη και πρέπει να αποφασίσουμε τα περί μακροαιρεσιμότητα. Είναι σαφής, σαφέστατη η εντολή που έχουμε. Δεν δεχόμαστε τη μακροαιρεσιμότητα. Δεν μπορούμε να δεχθούμε τη σχέση αυτή έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα. Ήδη Υπάρχει αρκετή νομοθεσία που έχει τεθεί σε ισχύ. Έχουμε τις έξι το 2 μετά. Άρα δεν χρειάζεται νομίζω αυτή με σχέση με τα περιφερειακά ταμεία να προχωρήσει. Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικότερα στοιχεία τα οποία είναι υποδιαπραγμάτευση. Τώρα, πρακτικά βλέπετε στον κατάλογο ακριβώς τι έχουμε συμφωνήσει, ποια σημαίνει υποδιαπραγμάτευση ακόμα και ποια δεν τα έχουμε ακόμη συζητήσει ή είναι τόσο δύσκολα που δεν είχαμε κάνει μια πλήρη ανταλλαγή απόψεων επ' αυτό. Τα τελευταία θέματα που σας ανέφερα ακριβώς σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται. Είμαι ανοιχτός να ακούσω τι ερωτήσεις σας σήμερα γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμα μία ή δύο συνεδριάσεις επιτροπής με σε αυτό το θέμα. Ε, και η Κωνσταντσε ίσως ε, είναι η ώρα να πάρει το μπαλάκι από μένα και να συνεχίσει. Πρόεδρος, δεν μαθαίνετε κύριε Φανίστελ Ρόι. Πρέπει να μου το πείτε και εγώ θα δώσω το λόγο στην Κωνσταντζή. Κωνσταντζή λοιπόν για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ε, ευγενική πρόσκληση. Δεν θα πω πολλά, γιατί ο Λάμπερτ ε, τα είπε τόσο ωραία. Αύριο θα γίνει ο τελευταίος, ε, από ό,τι φαίνεται, τριμερής διάλογος υπό Ιρλανδική Προεδρία και ελπίζω ότι θα είναι ένα σημαντικό βήμα πρόοδου, όχι μόνο για το κοινωνικό ταμείο, αλλά και για τις άλλες τέσσερις θεματικές κατηγορίες. Υπάρχει τώρα ήδη ένα σχέδιο έκθεσης για την ε, συζήτηση τον Ιούλιο, ένα προσωρινό σχέδιο. Εδώ φαίνεται ότι το Κοινοβούλιο επέτυχε τους ε, σημαντικούς στόχους του και ελπίζω ότι και αύριο θα επιτύχουμε αυτά που απομένουν να επιτευχθούν και θα καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό που θα μας επιτρέψει να υπάρχει ασφάλεια προγραμματισμού στις περιφέρειες για να συνεχιστούν τα επιχειρησιακά προγράμματα και να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τις ενέργειες των περιφερειών. Ξέρετε ότι έγιναν για τον γενικό κανονισμό 50 τριμερείς διάλογοι, κάπου έπρεπε να καταλήξουν. Μία παρατήρηση. Γιατί με ρώτησαν κάποιοι συνάδελφοι γι' αυτό. Οι διάφοροι κανονισμοί για τα διάφορα ταμεία σχετίζονται φυσικά με το γενικό κανονισμό και σε ορισμένα σημεία υπάρχουν ε, σαφείς επικαλύψεις. Ένα είναι απόλυτα σαφές. Εάν υπάρξουν ε, ασυνέπειες μεταξύ των διαφόρων κειμένων, το κείμενο αναφοράς θα είναι ο γενικός κανονισμός ή για θεματικές προτεραιότητες ή για οτιδήποτε Φυσικά βεβαίως ε, θα γίνει μετά εξέταση των κειμένων και γλωσσική εξέταση και όπως είπα ο γενικός κανονισμός θα ισχύει. Μην ανησυχείτε αν υπάρχουν δηλαδή κάποιες ασυνέπειες. Πάντα σε διαπραγματεύσεις, σε όλες τις διαπραγματεύσεις είπαμε ότι φυσικά θα πρέπει να ελέγξουμε και τα γλωσσικά θέματα, να υπάρχει παντού η ίδια διατύπωση Μην νομίζετε ότι θα έχουμε τέτοιου τύπου προβλήματα και θα χρειαστούν άλλες ε, τροπολογίες. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται τώρα να συζητήσω ένα-ένα τα ε, ε, μία-μία τις θεματικές κατηγορίες και να σας πω τι συμφωνήθηκε και τι είναι ακόμη ανοιχτό. Αλλά θα κάνω άλλη μία παρατήρηση. θα το πούμε και αύριο όταν θα αποφασίσουμε τα ποσοστά συγχρηματοδότησης. Δεν καταλαβαίνω γιατί τα κράτη-μέλη εμένουν σε ένα τόσο περίπλοκο σύστημα. Εμείς κάναμε μια πολύ απλή πρόταση που κατά τη γνώμη μας λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των περιφερειών πάρα πολύ καλά. Και ελπίζω αυτό το σημαντικό για τις περιφέρειες ε, σημείο να το διαπραγματευτούμε αύριο και να τα καταφέρουμε. Και είναι σαφέ και το λέει και η έκθεση τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων των τριών οργάνων, βεβαίω είναι συνήθω ε, συμβιβασμό. Σε ένα συμβασμό κανεί δεν είναι 100% ικανοποιημένο, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε γενικά ικανοποιημένοι. Αυτά που επιτύχαμε είναι σημαντικά. Αν δεν είχε υπάρξει συμφωνία με το Συμβούλιο, τότε είναι πολύ σημαντικό για μα να, να μην υπάρξει καμία περαιτέρω αλλαγή. Έχουμε την εντολή μας ή θα έχουμε στην έκθεση την άποψη του Κοινοβουλίου ή θα έχουμε το συμβιβασμό στον οποίο θα έχουν καταλήξει τα τρία όργανα. Οι προτάσεις που έχουν γίνει λοιπόν να υποβληθούν τροπολογίες ε, δεν έχουν έννοια. Ή θα υπάρχουν τροπολογίες που θα είναι κατά του συμβασμού που θα έχουμε επιτύχει ή θα είναι κατά τη θέση του Κοινοβουλίου και τη εντολή μα. Δεν έχουν έννοια λοιπόν. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Αλλά θεωρώ ότι τον Ιούλιο θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στην ψηφοφορία και θα πρέπει μετά οι συνάδελφοι να ενημερώσουν την κοινή γνώμη για αυτά που θα έχουμε επιτύχει το, θέμα δεν είναι μόνο να ψηφίζουμε με τους ε, πολυσέλιδους καταλόγους προφοριών, είναι να ενημερώνουμε και τους προφόρους μας, τις περιφέρειες, ε, ότι έχουμε επιτύχει σημαντικά πράγματα για τις περιφέρειες. Να αρκεστώ σε αυτά, αν υπάρχουν ε, συγκεκριμένες ερωτήσεις. Νομίζω ότι και ο Λάμπερτ και εγώ είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε πληροφόρηση, να απαντήσουμε για λεπτομέρειες και ευχαριστώ πολύ. Ο Γκουτμάνης δεν είναι παρόν. Η εκπρόσωπος των Πρασίνων. Δεν έχουμε φιλελευθέρους. Οπότε η εκπρόσωπος των Πρασίνων, αν θέλει το λόγο, τον έχει. Όχι, τίποτα. Υπόθηκαν όλα. Δεν είναι ευθύνη του Κοινοβουλίου ότι υπάρχει καθυστέρηση. Αυτό θέλω να τονίσω. Χρειαστήκαμε τρομερά πολύ χρόνο και είναι σαφές και είναι σαφές ότι είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα υπό την Ελλαδική Προεδρία παράλληλα με την Ολομέλεια τριμερείς διαλόγους γιατί θέλαμε να καταλήξουμε συμφωνία και για το θέμα του Κοινωνικού Ταμείου. Είχαμε προσεγγίσει πολύ για συμφωνία αλλά τελικά το Συμβούλιο δεν συμφώνησε. Και τώρα αυτή τη βδομάδα λέει το Συμβούλιο ξαφνικά θέλουμε νέο τριμερή διάλογο, θέλουμε συμφωνία. Είναι σαφές ότι άσκησε πίεση η Ιρλανδική Προεδρία στα κράτη-μέλη που θέλουν να υπάρχει ασφάλεια για τον προγραμματισμό. Νομίζω ότι δεν αξιοποίησε πλήρως την εντολή της η Ιρλανδική Προεδρία, δεν αξιοποίησε τις δυνατότητες που υπήρχαν να ε, διαπραγματευτούμε και να καταλήξουμε νωρίτερα υπήρχε χρόνος. Με ανυπομονησία ε, περιμένω να δω εάν θα έχουμε αποτέλεσμα. Όλοι χρειάζεται να αλλάξουμε τον προγραμματισμό μας για να δούμε, ε, να επιτρέψουμε να γίνει αυτή η συνάντηση αύριο. Ελπίζω να καταλήξουμε. Είπα, επαναλαμβάνω λοιπόν, δεν φταίμε εμεί, δεν φταίει η διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου φταίει η Ιρλανδική Προεδρία για την καθυστέρηση ενό εξαμήνου. Δεν ήταν διατεθειμένοι να διαπραγματευτούν. Αντίθετα με άλλε Προεδρίε. Συνήθω προσπαθούν οι Προεδρίε. Και έκαναν και γι' αυτό το θέμα προσπάθεια άλλε Προεδρίε. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω αυτό που είπε νωρίτερα ο Λάμπερτ στην εισαγωγή που μας έκανε το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι η δημιουργία αυτού του αποθεματικού επίδοσης για όλα τα ταμεία. 7% και μετά μακροοικονομική αρεσιμότητα για τη δυνατότητα μεταφοράς χρηματοδότησης, μεταφοράς πιστώσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων σε μια δεδομένη χώρα. Νομίζω ότι αυτά είναι τα μείζωνα ζητήματα θα ήθελα λοιπόν οι διαπραγματεύσεις να ολοκληρωθούν επιτυχώς. Αν έχει δίκιο η Κωνσταντσε και είναι πράγματι ο τελευταίος τριμερής διάλογος, θα είμαι πολύ ικανοποιημένος. Πρόεδρος, κάποιος την ο κύριος μαζί όχι, άρα κανείς. Ποιος άλλος θέλει να μιλήσει. Θέλετε μήπως ε, οι δύο συγκητές Λάμπερ Κωνσταντσε να απαντήσετε στο Σκιώδης. Όχι. Θα Λερόι. Μια λέξη να πω για το Συμβούλιο. υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις όπου επέδειξαν κάποια προθυμία, κάποια διάθεση να κινηθούν, αλλά ήταν ελάχιστες. Έπρεπε να τις περιμένουμε αυτές τις στιγμές και ξέρετε, μας κόστησε πολύ χρόνο αυτό, συμφωνώ. Yeah, but patient space also. We... Αποδίδει υπομονεό. Επιμένω νικά, ξέρετε, πολλές φορές. Η Κωνσταντσε. Μια φράση. Μια φράση για αυτή την Προεδρία. Δεν πάμε αύριο για να υπάρξει οπωσδήποτε συμφωνία. Θα επιχειρήσουμε να διαπραγματευτούμε για να καταλήξουμε σε καλό αποτέλεσμα. Δεν θέλουμε συμφωνία πάση θυσία. Δεν θέλουμε να πάμε λέγοντας εντάξει είναι ο τελευταίος ε, τριμερής διάλογος. Δεν είναι αυτός ο στόχος ε, των καθηκόντων μας. Γι' αυτό είμαι μεν συγκρατημένα αισιόδοξη Ελπίζω αύριο να τα καταφέρουμε να κλείσουν οι διαπραγματεύσει με ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά απόλυτα σίγουροι δυστυχώς δεν είμαι. Πρόεδρος. Τον Ιούλιο να είστε όλοι γιατί θα ψηφίσουμε. Σα υπενθυμίζω. Δεν έχω κάποιο σχόλιο προ το σημείο αυτό τη μεσικής διάταξη. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο σχέδιο έκθεση, έκθεση του Γιάνν Ολμπριχτ. Για το Βελγικό των Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα κάνω μια σύντομη παρουσίαση πιο πολύ θα σχολιάσω κάποιου πίνακε στη λογική του Συμβουλίου, τι επαγγελματικέ προτεραιότητε, την αστική διάσταση, θεματική συγκέντρωση κτλ. κτλ. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι είχαμε 13 τριμήρες διαλόγου και μια σειρά από τεχνικές συναντήσεις. Έχουμε επιτύχει συμφωνία μέχρι σήμερα για το σύνολο των διατάξεων. Ουσιαστικά έχουμε ολοκληρώσει δηλαδή Υπάρχουν κάποια, κάποιες ελλείψεις, όχι ως προς ε, τα σημεία των οποίων έχουμε συμφωνήσει, αλλά για την αριστικοποίηση ε, του τελικού κειμένου. Λόγω της συμφωνίας ε, και για το κοινωνικό ταμείο και επειδή θα επηρεαστεί το θέμα της θεματικής συγκέντρωσης λόγω του CPR, Θέλουμε να κάνουμε τη διατύπωση να είναι προσαρμοσμένη σε αυτές τις νέες εξελίξεις και για τις, ε, και τις περιφέρειες, είχαμε ένα ζήτημα και όχι όσον αφορά τη χρηματοδότηση αλλά τη βοήθεια. Περιέργως αυτό ήταν το πιο εκρηκτικό θέμα. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διαπραγμάτευση ε, νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου Οικονομικής ε, Υπηρεσίας του, της Κομισιόν ε, τελικά κατάφεραν να συμφωνήσουν. Και έχετε και τις προτάσεις αυτές με τη μορφή τροπολογίας που καταθέτει ο εισηγητής. Σε ό,τι αφορά τώρα τα βασικά σημεία της συμφωνίας, τα συγκεκριμένα κεφάλαια, σε ό,τι αφορά την υποστήριξη. Θα σας θυμίσω ότι υπήρχαν κάποια δύσκολα σημεία για τα οποία όμως βρήκαμε λύση. Και ποια ήταν αυτά. Πρώτον, μεγάλες επιχειρήσεις ε, και παραγωγικές επενδύσεις. Εμείς συμφωνήσαμε, οπότε στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας ε, και για τη μετάβαση σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών. Ε, θέλουμε λοιπόν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν μέσα, γιατί ήταν ένα επίμαχο θέμα. Καταφέραμε επίσης ως Κοινοβούλιο να μπουν οι μικρές τουριστικές ε, υποδομές μικρής κλίμακας. Συμφωνήσαμε να διαγραφεί η απαγόρευση επενδύσεων σε τομείς διάφορους όπως είναι ο τουρισμός ή τη τεχνολογία προφορών επικοινωνιών ε, σε κάποιες περιφέρειες. Γιατί δεν θα μπορούσε να ισχύσει ε, στο πλαίσιο του κανονισμού. Και επίσης έχουμε μια απαγόρευση, πιο σημαντικό αυτό, στις αεροπορικές υποδομές οι επενδύσεις, εάν δεν ε, επιτρέπουν την περιβαλλοντική προστασία, απαγορεύονται. Και ισχύει αυτό όχι μόνο για το ΕΤΠΑ, είναι σημαντικό για τις επενδύσεις ΕΤΠΑ στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Θα είναι δυνατό λοιπόν να γίνονται επενδύσεις σε ευρωπαϊκές υποδομές, αλλά πάντοτε σε σχέση με την περιβαλλοντική προστασία, αν υπάρχει αυτή η παράμετρος. Για τις προτεραιότητες τώρα επενδύσεων. Υπάρχουν κάποια σημεία για τα οποία επέδειξε ιδιαίτερα προθυμία ναι, Κομισιόν. και αυτό μας εξέπληξε. Για παράδειγμα, η οικολογική καινοτομία. Εμείς καταφέραμε την οικολογική καινοτομία να τη συμπεριλάβουμε ε, και επίσης ε, τις δημιουργικές ε, βιομηχανίες και πολιτιστικές, τον πολιτιστικό κλάδο. Αυτό θα το δείτε στις τροπολογίες. Επίσης η culture στι αιτιολογικέ σκέψει θα δείτε ακριβώ πώ εννοούμε τα πράγματα και με ζωντανά των δαπανών. Επίση, θα μπορούμε να ε, χρηματοδοτήσουμε επενδύσει ε, σε μικρομεσαίε επιχειρήσει για την ανάπτυξη πρώτων και υπηρεσιών, για παράδειγμα. Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση τώρα. Όχι για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, μιλάμε για όλε τι επιχειρήσει και για τι μεγάλε Η επιλεξιμότητα για δαπάνες ε, με στόχο ενεργειακή απόδοση. Το θεματική στόχη. Η αστική κινητικότητα είναι πλέον και αυτή προτεραιότητα μέσα στο στόχο μας για χαμηλές εκπομπές. καταφέραμε να πετύχουμε επίσης την πρόθεση τεχνολογιών ε, χαμηλών εκπομπών, ή ενέργεια και άλλες μορφές ενέργειας, αλλά και να τονίσουμε το, την προσέγγιση ε, οικοσύστημα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και επιλεξιμότητα ε, για επενδύσεις στον τομέα του ύδατος και των αποβλήτων. Πολύ σημαντικό. Ξεπερνάμε την προσαρμογή στο κοινωτικό κεκτημένο. Αυτό ήταν ε, επίμαχο ζήτημα, αν δηλαδή μπορούμε να ξεπεράσουμε ή όχι αυτή ε, την προσαρμογή του κοινωτικού κεκτημένου, θα δείτε τα σχετικά και στη συζήτηση για τις κρατικές ενισχύσεις, αν ε, μπορούμε δηλαδή να πάμε πιο πέρα από το κοινωτικό κεκτημένο. Επίσης για την βελτίωση αστικού περιβάλλοντος, την αναζωγόνηση των πόλεων ή κάποιες ε, περιοχές οι οποίες αναπλάστηκαν, συμπεριελήφθησαν όλα αυτά στην επιλεξιμότητα για επενδύσεις. Επίσης, ατμοσφαιρική ρήπανση, ρήπανση, ελήφθησαν υπόψη. Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για την ε, αποτελεσματικότητα των πόρων και ανάπτυξη όχι μόνο σιδηροδρομικών αλλά και αποκατάσταση σιδηροδρομικών συστημάτων. Πολύ ευρύτερε ε, λοιπόν δυνατότητε ε, για δαπάνε των κονδύλιων του ΕΤΠΑ. Επίση, για την πρόθεση μέτρων μείωση του ορίου στον των μεταφορών. Και εδώ προωθήσαμε την επιλεξιμότητα. Για ευφυή, e, διανομή, ε, αποθήκευση ενέργειας, παραγωγή ενέργειας. ενδογενές δυναμικό. Κάτι άλλο επίμαχο, θα το βρείτε όμως εδώ, ήταν κοινωνικές, ε, ψυχαγωγικές ε, και πολιτισμικές υπηρεσίες. Ψυχαγωγικές με ποια είναι, για να περιοριστεί ε, ο κοινωνικός αποκλεισμός και να προωθηθεί κοινωνική ένταξη. Κοινωνική αποκατάσταση μειονεκτικών περιοχών ή ομάδων επίσης ήταν ένα θέμα και ένα άλλο στοιχείο σε ό,τι αφορά την τελική συμφωνία που ελπίζουμε και να μην αλλάξει μετά τα συμπεράσματα του ΕΣΕΦ είναι πρώτον θα έχουμε τη συγκέντρωση σε τέσσερα τομείς means that uh, Είχαμε κάποια διαφωνία με το Συμβούλιο. Πρότεινε να είναι μία τουλάχιστον κατηγορία στις προτεραιότητες του Συμβούλου. Εμείς προτείναμε δύο. Η αρχική πρόταση της Κομισιόν ήταν τρεις, αλλά α, θεώρησε ότι είναι ακραία η πρόταση αυτή το Συμβούλιο και την απέρριψε, ενώ εμείς την υπερασπιστήκαμε στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων θέλαμε να υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση. Δύο τουλάχιστον από το 1, 3, 4. Τους τέσσερα. Τα τέσσερα θεματικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, χαμηλός, ε, χαμηλές εκπομπές και άλλα. Επίσης, θα, στόχος μας είναι η ενεργειακή απόδοση, ε, χαμηλές εκπομπές δεν είναι το ίδιο, αλλά τα χρησιμοποιούμε μαζί. Τουλάχιστον 20% του ΕΤΠΑ θα πάει εδώ, για τις πιο ανεπτυγμένες περιοχές. Τουλάχιστον 15% για τις περιοχές μετάβασης και τουλάχιστον 12% για τις λιγότερο ανεπτυγμένες ε, περιοχές. Αλλά, αν συμπεριληφθεί και το Ταμείο Συνοχής, θα είναι τουλάχιστον 15%. Εξαιρέσεις. ο μηχανισμός ε, αποζημιώσεων μεταξύ περιφερειών που μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη, δηλαδή επανεξορρόπηση για να, λάβουν, ε, για να είναι ίδιο το ποσοστό χρηματοδότηση όλων των περιφερειών. Πολύ επίμαχο το θέμα αυτό και μερικοί συνάδελφοι της Επιτροπής μας ε, επίσης τους ενδιαφέρει το ΝΑΤΣ 2, τα νησιά. Ε, αντιμετωπίζονται ως ε, λιγότερο ε, ανεπτυγμένες περιοχές. Μόνο και μόνο επειδή είναι νησιά. Είπαμε όλα τα νησιά να είναι στο ΝΑΤΣ 2, αλλά το Συμβούλιο διαφωνούσε κάθετα. Και επίσης και η Επιτροπή. Τελικά, τα περισσότερα από τα νησιά ΝΑΤΣ 2 θεωρούνται ως λιγότερο ανεπτυγμένα. Εκτός από τέσσερα. Βαλεαρίδες, Σαρδινία, Κορσική και κάποιο βόρειο νησί. Άλαντ. Άλλαντ. Γιατί δεν είναι και τόσο υπανάπτυκτες περιοχές. Προσπαθούμε να αποφασίζουμε με αντικειμενικά κριτήρια. για να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Είναι θέμα επανακάτικο. Τώρα είναι περιοχές που σταδιακά ε, βγαίνουν από τη χρηματοδότηση. Ε, αντιμετωπίζονται ως περιοχές περιφέρειες μετάβασης. Ε, ορισμένες είναι στη Γερμανία. Όχι θεματική συγκέντρωση για τις ε, εξόχως απομακρυσμένες περιοχές. Και εδώ υπήρξε μεγάλη σύγκρουση. και θα είναι διαφορετική η χρηματοδότηση των αεροκατοικημένων περιοχών. Εδώ είναι η εξαίρεση. Αστική διάσταση. Το περίφημο 5% του ΕΤΠΑ στα κράτη-μέλη. Θα δοθεί για πιλωτικά προγράμματα για βιώσιμες αστικές δράσεις. Και στις συμφωνίες εταιρική ε, σχέσης τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δουν πώς θα, να συμφωνήσουν πώς θα τα κατανείμουν. Ε, αυτό θα αφορά λοιπόν τις πόλεις και τα προάστια. Και θα πρέπει να δούμε σε ποιο επίπεδο θα παίρνονται οι αποφάσεις. Δεν συμφωνούσε το Συμβούλιο να λαμβάνονται αποφάσεις σε υψηλότερο επίπεδο. Κάποια κράτη-μέλη δεν το θέλουν αυτό. Άρα υπάρχει μια κλιμάκωση ανάλογα με το μέγεθος των προγραμμάτων, ποιο επίπεδο απόφαση, σε ποιο επίπεδο θα παίρνονται οι αποφάσεις. Θυμάστε και μια προηγούμενη φορά δεν έγινε δεκτή μια παρόμοια πρόταση. Στην προηγούμενη θητεία. Τώρα κάτι επιτύχαμε. 5% λοιπόν για βιώσιμες ε, αστικές δράσεις. όχι μόνο μέσω ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων, αλλά και με συγκεκριμένα προγράμματα, ειδικά, μπορούν να αξιοποιήσουν ε, λοιπόν τα κράτη-μέλη αυτό το 5% είτε συνολικά μέσω ενός προγράμματος είτε κατά τμήματα. Δεν υπάρχει κατάλογος των πόλεων στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης, αλλά θα υπάρχει ένας κατάλογος κριτηρίων. Και δεν θα υπάρξει πλατφόρμα αστικής ανάπτυξης για 300 πόλεις, αλλά ένα δίκτυο αστικής ανάπτυξης. Δεν είναι απλώς αλλαγή διατύπωσης. Είναι ουσιώδης αλλαγή. γιατί έκανε μια μελέτη η Επιτροπή για να δει πώς λειτουργεί αυτό το μέσο. ...2,02% του ΕΤΠΑ θα δοθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για καινοτόμες δράσεις. Θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, διαγωνισμούς. Δεν θα αλλάξουν λοιπόν ε, τα πράγματα για τις ε, καινοτόμες δράσεις 330 εκατομμύρια. Το μόνο στοιχείο όπου στα συμπεράσματα του Συμβουλίου υπήρχε συγκεκριμένο ποσό. Όπως και στους άλλους κανονισμούς, υπάρχει το θέμα των δικτών απόδοσης. θα υπάρχει δυνατότητα ε, μέσω κατεξοδότηση πράξεων να αλλάζουν αυτά. Δεν θα υπάρξει τώρα τροποποίηση. Αλλά θα είναι δυνατόν ε, μέσω κατεξοδότηση πράξεων να τροποποιήσουμε αργότερα. Ο κατάλογος των δικτών θα βασιστεί στην πρόταση του Συμβουλίου που είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας ε, μελετών και διαβούλευσης διετή. Δεν χρειάζεται λοιπόν να αλλάξουν οι δείκτες. Ένα από το πιο δύσκολο πρόβλημα είναι πώς θα λειτουργήσει η βοήθεια. Η γενική πρόθεση της εντολής μας ήταν να απλουστευτεί η κατάσταση για τις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές, να μην υπάρχουν περισσότερα εμπόδια. Να μην τους υποχρεώνουμε να δίνουν, για παράδειγμα, ειδική ειδοποίηση γιατί η κατάστασή τους είναι ιδιαίτερη. Και ελπίζω το τελικό κείμενο να επιτρέψει απλές διατάξεις. Θα δείτε επίσης ότι αναφέρομαι στα στοιχεία του διαχείρισης κινδύνου, βιώσιμος τουρισμός, ε, πολιτισμός και πολιτιστική κληρονομιά, καθορισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ε, υπηρεσίες που βασίζονται στην κοινότητα. Για όλα αυτά τα θέματα είπαμε ότι θα συμπεριληφθούν, αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε στη διατύπωση. Είπαμε ότι θα συμπεριληφθούν σε αιτιολογικές σκέψεις. Δεν το συζητήσαμε στις διαπραγματεύσεις. Όπως βλέπετε, ενώ είναι σύντομος ο κανονισμός, υπάρχουν πολλά σημαντικά στοιχεία για όσους μετά θα πρέπει να τον εφαρμόσουν Ευχαριστώ λοιπόν την διαπραγματευτική ομάδα για την ε, διάθεση συμβασμών που επέδειξε. Υπήρξαν βέβαια δυσχέρειες, αλλά είχαμε ε, μια πολύ ειλικρινή διάθεση ακόμη και να διαφωνήσουμε αλλά με επικοδομητικό τρόπο. Δεν ήμασταν πάντα βέβαια ε, όλοι πολύ ευγενείς και γι' αυτό πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Είναι πρόβλημα του εισηγητή αυτό. Ελπίζω λοιπόν τον Ιούλιο να είμαστε έτοιμοι. Θέλουμε να αποστείλουμε προς τις περιφέρειες το μήνυμα ότι εμείς είμαστε έτοιμοι και ελπίζουμε και το Συμβούλιο να επιδείξει θετική στάση. Θα ξεκινήσω με τους σκιώδεις. Ευχαριστώ. Ή μίλησα ήδη την προηγούμενη φορά για τα αποτελέσματα και τους και αυτά τα οποία έχουν, ε, είχαν τότε παραμείνει ανοιχτά έχουν έκτοτε και με βάση την εντολή μας είχαμε εντολή με την οποία ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσει και το πνεύμα της εντολής το τηρήσαμε. Φυσικά δεν μπορούμε να τα επιτύχουμε ποτέ όλα, αλλά νομίζω ότι τηρήσαμε τη βασική μας γραμμή και επιτύχαμε να περάσει. Θα θέλαμε να έχουμε επιτύχει περισσότερα βεβαίως, αλλά ε, εμείς από την Επιτροπή μας είμαστε μόνο ένα τμήμα της διαπραγμάτευσης, υπάρχουν και άλλοι. Νομίζω λοιπόν ότι πολλές περιφέρειες θα θεωρήσουν πολύ ικανοποιητικό αυτό το αποτέλεσμα του τετάρτου στόχου δηλαδή που επιτύχαμε. Όπως είπε Γιάννη, ήταν σημαντικό να ε, υποστηρίξουμε όχι μόνο τις μικρομεσαίες αλλά ακόμη και μεγάλες επιχειρήσεις που λειτουργούν σε διάφορες περιφέρειες και επίσης χαίρομαι, χαίρομαι που και οι πόλεις μπόρεσαν να βάλουν το πόδι στην ε, πόρτα ναι ε, δεν επιτύχαμε όσα θα θέλαμε για τις πόλεις αλλά βάλαμε το πόδι στην πόρτα επίσης η προώθηση του πολιτισμού και του αθλητισμού υπήρχε ένας Αυστριακός συνάδελφος που είπε πόσες θέσεις εργασίας δημιουργούν αυτοί οι τομείς. Σημαντικό που επιβάλαμε και εδώ την άποψή μας. Όπως είπε και ο Γιάνν, όσα επιτύχαμε ε, οφείλονται και στον τρόπο με τον οποίο διαπραγματευθήκαμε. Υπήρχε μια κάποια ενότητα, αλλά έπαιξε ρόλο και η ηγεσία της διαπραγματευτικής μας, της διαπραγματευτικής μας ομάδα, ομάδας είναι σημαντικό να επιτυγχάνεται η ενότητα μεταξύ της διαπραγματευτικής μας ομάδας γιατί αν υπάρχουν διαφωνίες τότε ευκολότερα ε, επιτυχάνουν οι αντίπαλοι μας να περάσει η δική τους άποψη. Ευχαριστώ λοιπόν τους πάντες, ευχαριστώ τον Προεδρεύοντα της διαπραγματευτικής ομάδας, θαυμάσια εργασία και όπως είπα τηρήσαμε το πνεύμα της εντολής. Ε, δεν τα επιτύχαμε όλα αλλά θα έχουμε και επόμενες διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Η Ρέικα δεν είναι εδώ. Καρίμ δεν είναι εδώ. Κύριε Βλάσακ, θέλετε το λόγο. Νομίζω ότι όλα τα είπε ο Ιαν. Ε, να τον ευχαριστήσω αυτόν και την ομάδα του για τη συμβιβαστική πρόταση. Νομίζω ότι τα βασικά θέματα καλύφθηκαν και οι μεγάλες επιχειρήσεις θα υποστηρίζονται όπως και οι μεσαίες και οι μικρές. Και θα υπάρξει στήριξη επίσης και για τον πολιτισμό και για τον αθλητισμό. Ευχαριστώ. Η Κορνέλια. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Ο οποίος χρειάστηκε να ε, διαφωνήσει και με το Συμβούλιο και με μερικούς εξημών, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται. Παρ' όλα αυτά, το πνεύμα ήταν θετικό στην διαπραγματευτική ομάδα. Νομίζω ότι υπερασπιστήκαμε τις θέσεις μας. Το πεδίο εφαρμογής για τις μικρομεσαίες, αυτό είναι σημαντικό. Είπαμε ότι και μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει να μπορούν να ληφθούν υπόψη. εφόσον κάνουν κάτι ανάλογο με τις μικρομεσαίες, προτεραιότητα τις επενδύσεις. Με εξενέβρισε ότι δεν τα καταφέραμε με τις περιθωριοποιημένες κοινότητες. Είναι στις αιτολογικές σκέψεις βεβαίως. Καλύτερα θα ήταν να υπάρχει σε ένα άρθρο του κειμένου θεματική στόχη. Ξέρετε δεν ε, υπήρχε και μεγάλος ενθουσιασμός γι' αυτό, για μας, γιατί ως ομάδα θεωρούμε ότι περιορίζει, περιορίζει τον τρόπο εφαρμογής. Δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνουν. Θα δούμε βέβαια εάν αυτά τα οποία ε, επιτύχαμε θα εφαρμοστούν με τρόπο μη γραφειοκρατικό. Αλλά αυτό θα φανεί κατόπιν κατά την εφαρμογή. Θέματα περιβάλλοντος τα συζητήσαμε εντονότατα. Εδώ έγιναν οι μεγάλες ε, αντιπαραθέσεις. Δεν ξέρω αν συμφωνώ με αυτό που επιτεύχθηκε για τα ε, αεροδρόμια και για τις ευφυείς μορφές ενέργειας, αλλά τουλάχιστον αποφύγαμε τα χειρότερα για τις ε, πιο απομακρυσμένες περιοχέ και τα νησιά δεν είμαι τόσο ικανοποιημένη. Αλλά, εν για την σταδιακή κατάργηση, phasing out, είναι οι περιοχές μετάβασης. Πρόκειται λοιπόν για το 15%. Δεν μας ικανοποιεί τόσο πολύ η κατάσταση. Θα θέλαμε να έχουν αυξηθεί αυτά τα όρια. Αλλά κατά τα άλλα, δώσαμε καλές μάχες. Και σας συγχαίρω γι' αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στον συνάδελφο Όλμπριτς. Θα ήθελα να εκφράσω και την απογοήτευσή μου όμως σε σχέση με τα αποτελέσματα στο οποίο καταλήγουμε. Εμεί από τη μία προωθούμε την αντίληψη για την εδαφική συνοχή, για την περιφερειακή πολιτική και βρισκόμαστε απέναντι στη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία είναι συγκεντρωτική, ξεπερασμένη. Είναι κάτι το οποίο έχει σαν βασικό στόχο τη διατήρηση της καθεστικής τάξης. Εμείς προσπαθούμε δηλαδή για να ξεπεράσουμε την δυσφορία την οικονομική που πνίγει ιδιαίτερα τις περιφέρειές μας. Βλέπουμε όμως τους γενικούς στόχους τους οποίους θέτει η πολιτική 2020 Απ' την άλλη όμως βλέπουμε ότι εμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διατήρηση του status quo. Οπότε θα πρέπει εμείς να ενισχύσουμε τη δική μας θέση και τους εισηγητές μας. Και δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε γιατί αλλιώς θα χάσουμε άλλα 7 χρόνια όπου η απόσταση από την περιφέρεια στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αυξάνεται οι ταχύτητες οικονομικής ανάπτυξης θα είναι μικρότερες, η φτώχεια θα είναι μεγαλύτερη και θα υπάρχει και η υπανάπτυξη. Να μιλήσω τώρα για τον νησιωτικό χαρακτήρα. Επανειλημμένα σε αυτό το κοινοβούλιο και τον προηγούμενο Ιούλιο ε, για την περιφέρεια της Μεσογείου είπαμε ότι ε, ο ε, νησιωτικός χαρακτήρας είναι ένα μειονέκτημα, όχι όμως σε σχέση με το ΑΕΠ. Δεν μπορούμε εμείς τώρα να δεχτούμε την κατοδοριοποίηση των ίσων σε α, β κτλ. Ίσως το ΑΕΠ των Βαλεαρίων Ίσων ή η Σαρδινία να έχουν ένα ΑΕΠ και το γνωρίζω αυτό από την παρουσία ενός δηληστηρίου το οποίο πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή αλλά αυτό δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία σε σχέση με τα έσοδα του τοπικού πληθυσμού και θα πρέπει να εξαιρεθεί η Σαρδινία. Όχι, ο νησιωτικός χαρακτήρας μας εξαιρεί, μας αποκλεί από την ενιαία αγορά, από τη συνέχεια των οδικών μεταφορών. Μια ολόκληρη σειρά μειονεκτημάτων και θα πρέπει εμείς χωρίς καμία εξαίρεση να συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα νησιά επανέρχομαι, θα πρέπει μέχρι τέλους να παλεύουμε, εγώ και η πολιτική μου ομάδα, θα δώσουμε τη μάχη αυτή, μαζί και με άλλες μάχες βέβαια, τις οποίες δεν αναφέρω τώρα γιατί δεν έχω χρόνο, αλλά θα πρέπει να εμείνουμε στις θέσεις μας, γιατί αλλιώς η απόσταση κέντρου-περιφέρειας θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο και αυτό είναι καταδικαστέο. Φραντσέσκα Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ πλήρως με τον προλαλήσαντα, τον κύριο Ούτζιας. Καταλαβαίνει κανείς ότι από τα αποτελέσματα στα οποία έχουμε καταλήξει και τα οποία ακούσαμε εδώ σήμερα, σίγουρα έχει, γίνει, έχει προηγηθεί μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά, σίγουρα πάρα πολλά στοιχεία έχουν προωθηθεί και ήταν θετικά, διαπιστώνουμε την προσπάθεια του εισηγητή, μια προσπάθεια απέναντι στην επικυριαρχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά αυτό ακριβώς δεν επιτρέπει να προωθήσουμε όλες τις θέσεις μας, εμάς σαν Κοινοβούλιο και σαν Επιτροπή Περιφερικής Ανάπτυξης. Είμαι νέα βέβαια στην Επιτροπή σας, αλλά το αναγνωρίζω αυτό. Τους τελευταίους μήνες προσπάθησα να κατανοήσω σε βάθος αυτά τα οποία Eh, Να κατανοήσουμε λοιπόν ποιοι είναι οι πολιτικοί στόχοι τους οποίους θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 στον τομέα της εδαφικής συνοχής και σε μια προσπάθεια ακόμα πιο μεγάλη για τη σμίκρινση των διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλές φορές μέσα στις περιφέρειες των χωρών σε κάθε χώρα. Έμαθα λοιπόν και εγώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσπαθήσει να προωθήσει τις πολιτικές της αρχές και προσπάθησε αυτά να τα συνοδεύσει με συγκεκριμένα μέτρα τα οποία να είναι συνεκτικά με την πολιτική της. Υπήρξαν βέβαια αντιστάσεις προφανής από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διαψεύδουν τους πολιτικούς μας στόχους. Διαψεύδουν αυτούς τους στόχους που είναι απαραίτητοι για να μπορέσει κανείς ε, να καταλήξει σε αυτό το τόσο επιθυμητό ομοιογενές και μακροπρόθεσμο στάδιο ανάπτυξης. Γι' αυτό λοιπόν οφείλω να υπογραμμίσω ότι ιδιαίτερα για το θέμα του νησιωτικού χαρακτήρα ναι μεν υπάρχει ένα μικρό βήμα αλλά πολύ φοβάμαι ότι μετά γίνονται δύο βήματα προς τα πίσω όσο ξεκαθαρίζονται οι θέσεις και όσο ακριβώς κατανοούμε το τι συμβαίνει. Τώρα για τη θεματολογική συγκέντρωση. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια αντίφαση η οποία πρέπει να ξεπεραστεί. Υπάρχει μια σαφής ε, διάκριση περαιτέρω ανάμεσα σε εδάφη, σε περιφέρειες οι οποίες έτσι κι αλλιώς αντιμετωπίζονται αρνητικά σε σχέση με άλλες και αν δεν κατάλαβα καλά, παρά το κείμενο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας, οι περιοχές ΝΑΤΣ 2, οι νησιωτικές περιοχές, έχουν τη δυνατότητα απόκλησης από τις βασικές αρχές της θεματολογικής συγκέντρωσης. Παρ' όλα αυτά κάποιες νησιωτικές περιοχές και εδώ θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε με ποιο τρόπο γίνεται η εξαίρεση αυτή και πώς ακριβώς θα επιλέγονται τα νησιά τα οποία θα εξαιρούνται και αναφέρομαι εδώ πάντα σε νησιά σαν τη Σαρδινία Υπάρχει μια διάκριση, ένας αποκλισμός, ο οποίος δεν είναι κατανοητός από καμία μα καμία άποψη. Θα πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε το θέμα του τρόπου υπολογισμού της ανάπτυξης των περιοχών αυτών των νησιών με βάση το τοπικό ΑΕΠ σίγουρα είναι ένας δείκτης από τους πιο απλούς και εύχριστος για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε νομοθετικές προτάσεις και να δώσουμε κίνητρα για την ανάπτυξη των περιφερειών. Αλλά όπως είπε και ο συνάλφος Ουτζίας πριν, και αναφέρομαι στη Σαρδινία την οποία γνωρίζω καλά, ο δείκτης αυτός του ΑΕΠ ε, αντιπροσωπεύει θα έλεγα μια ειδική κατάσταση στη Σαρδινία η οποία είναι απολύτως στρεβλή. Τα στοιχεία αυτά για τα έσοδα τα οποία έχει είναι άνω του 75% του ευρωπαϊκού μέσου όρου μόνο και μόνο επειδή υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο δηληστήριο στο νότο του νησιού το οποίο αυξάνει τους αριθμούς αλλά το πόσο αυτό ωφελεί την οικονομία του νησιού είναι προφανές ότι δεν υπάρχουν ωφέλη. Παραμένουν λοιπόν πολλές καθυστερήσεις, παραμένουν πάρα πολλές διακρίσεις, παραμένουν πάρα πολλές αδικίες για τους πληθυσμούς των νησιωτικών περιοχών και γι' αυτό απαιτείται να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες απόκλησης εξαίρεσης έτσι ώστε ε, να υπάρξει μια ισότητα δυνατοτήτων τουλάχιστον, ισότητα ευκαιριών, η οποία να μπορεί να στηριχθεί και από τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε. Αλλιώς είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας σαν βουλευτές να προσπαθούμε να ασκήσουμε την πολιτική μας, να προσπαθούμε να φέρουμε τους πολίτες κοντά στην Ευρώπη, να προσπαθούμε να πείσουμε τις τοπικές αυτοδιοικήσεις για τη σημασία της Ευρώπης, κάτι το οποίο θα θέλαμε να κάνουμε σε καθημερινή βάση. Εστάρας. Ευχαριστώ πολύ. Στο ίδιο πνεύμα με αυτά που είπε ο εισηγητής, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω να συγχαρώ καταρχάς για το δουλειά του. Βέβαια γνωρίζετε ότι κατάγομαι από τις Βαλαρίδες και μαζί με τον συνάδελφο Ουτσίας και την σύντροφο από τη Σαρδινία σε όλες τις επιτροπές, πολλές και διάφορες που προασπίζονται τα νησιά, πραγματικά εκπλησόμαστε βλέποντας ιδίως για τις Βαλεαρίδες, την Κορσική και τη Σαρδινία τη διάκριση, τη διακριτική μεταχείριση έχουμε τα κονδύλια διασυνοριακής συνεργασίας. Δεν θέλει η Κομισιόν το Συμβούλιο αυτή τη μέγιστη απόσταση να την εξαλείψει. Δεν μπορούμε να ε, εκμεταλλευτούμε τα κονδύλια και ακόμη πάνω σε αυτό σε ό,τι αφορά την ευελιξία των θεματικών στόχων, μα ε, εξαιρούν από την εξαίρεση. Όλα τα νησιά μπορούν να έχουν ευελιξία ε, στο πλαίσιο τη θεματική συγκέντρωση πλην των τριών αυτών που σα ανέφερα και δεν μα εξηγεί κανεί το λόγο. Δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια. Ε, και για τι Βαλεαρίδε που έχουμε και το μεγαλύτερα, τα υψηλότερα ποσοστά εγκατάλειψη του σχολείου και τα υψηλότερα ποσοστά ενεργεία στην Ένωση. Με τι κριτήριο, με τι κριτήριο λοιπόν εμεί και τα άλλα νησιά μένουν εκτό. Ένα από τα επιτεύγματα της συνθήκης της Λισαβόνας είναι ο νησιωτικός χαρακτήρας άνευτια ε, διαφοράς και ε, να πρέπει κάπως να λαμβάνεται υπόψη. Ε, και θέλουμε και την εδαφική συνοχή. Μέχρι τώρα μιλάμε για την οικονομική και την κοινωνική συνοχή, όχι για την εδαφική. Στην Επιτροπή των Περιφερειών, στα Intergroups, εδώ έχουμε κάνει συζητήσει, έχουμε καταρτήσει εκθέσει, όλα αυτά τα τελευταία 20 χρόνια. Αν δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια, ε, ξημέρωσαν, ε, ξημέρωσε μια μέρα πριν από λίγες ε, μέρες για να δούμε ότι για άλλους ισχύουν κριτήρια, για άλλους όχι. Και είναι σαν να φτιάχνει το Συμβούλιο ένα κοστούμι για την κάθε περιφέρεια, για την κάθε χώρα. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται μετά. Πίσω από ε, το κάθε άνθρωπο είναι σαν να είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, συγκεκριμένα μάτια, μπορώ να το πω έτσι. Και για τα τρία αυτά νησιά έχουν εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει τίποτα. Εμείς λοιπόν όσοι πληττόμεθα και ενδιαφερόμαστε με αυτό, ε, από αυτό έχουμε ενώ στις δυνάμεις μας παρακαλώ όλους τους προσώπους ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να φροντίσετε να διορθωθεί η αδική αυτή που ούτε σωστή είναι ούτε και εξηγείται με κάποιο τρόπο. Αν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια μπορούμε να δεχτούμε κάποια πράγματα, αλλά να υπάρχει διάκριση γιατί κάποιου του ήρθε να βγάλει έξω κάποια νησιά ε, και τελικά να εφαρμοστούν επιχειρήματα που δεν είναι τα ίδια για όλους. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, ο Φρανσό Αλφονσί και μετά θα ρωτήσουμε την Κομισιόν για τα αντικειμενικά αυτά κριτήρια για τα νησιά. Ο Φρανσό Αλφονσί. Ε, να μιλήσει και η φωνή της Κορσικής ε, υπέρ ε, των νησιών, Βαλεαρίδες και Σαρδίνια μίλησαν και για το Άλλαντ. Το 174 από τις συνθήκη αφορά τις μειονεκτούσες ε, περιφέρειες. Μέχρι σήμερα οι αεροκατοικημένες και οι ορεινές περιοχές με τον ένα τον άλλο τρόπο μέσω του ΦΕΑΝΤΕ ε, ιδίως οι ορεινές περιοχές ε, ελήφθησαν υπόψη επειδή έχουν ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Δεν κατάλαβα να γίνεται εξαίρεση για τις ορεινές πάρα πολύ πλούσιες αυστριακές περιφέρειες που λειτουργούν όπως ε, οι άλλες ορεινές και στο πλαίσιο του ταμείου αυτού που σας προανέφερα λαμβάνουν τις ίδιες ενισχύσεις. Μήπως θέλει που είναι αυστριακός επίτροπος, δεν το ξέρω. Αλλά όταν βλέπουμε τεράστιες αναπτυξιακές διαφορές, τι γίνεται με τα νησιά. Έχουμε κάποιες διατάξεις, το 174 που σας προανέφερα. Ο στόχος είναι ε, να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες ε, ενός εδάφους σε σχέση με τα μειονεκτήματα. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες των νησιών, είναι ότι από οικονομική πλευρά είναι ευάλωτα τα νησιά ε, όταν έχουμε μια αρνητική συγκυρία, ιδίω ε, στην περίπτωση των Βαλεαρίδων, με πολύ μεγάλη σημασία της τουριστικής σα. Πρέπει λοιπόν ε, να αντιδράσουμε όταν έχουμε προσταθεροποίηση της μικροοικονομίας καιρό κρίση. Και από την άλλη πλευρά πρέπει να αντιμετωπίσουμε ανάγκε εξοπλισμού, που είναι τελείω διαφορετικέ σε ένα νησί, υποδομές πρόσβασης, για τη διάθεση στο εμπόριο, για την πρόσβαση στο ε, εμπόριο στην νέα αγορά. Είναι άλλε συνδομέ. Θα πρέπει επίση το κόστο διαβίωση λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα να ληφθεί υπόψη. Όλα αυτά είναι ευαισθησίε, είναι ιδιαιτερότητε, πολύ σημαντικέ. Το πνεύμα τη συνθήκη νομίζω είναι και για τα νησιά και για τα βουνά να προωθήσει διατάξει οποίε θα ισχύουν και θα εφαρμόζονται ομοιόμορφα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ, ο Γιάννη. Α, με συγχωρείτε πολύ. Θέλω να μιλήσει και η κυρία Κρέλ. Entschuldigung, äh, Με συγχωρείτε που μπαίνω μέσα στο, στη συζήτηση για το δικό σου κανονισμό. Ήθελα να σας πω να, να διευκρινίσω ότι στη Γερμανία και στην Αυστρία όλες οι ορεινές περιοχές ε, αποφασίζεται πώς θα αντιμετωπιστούν ε, και με βάση τα κριτήρια παίρνουν, ε, επειδή θεωρούνται πολύ αναπτυγμένες περιοχές, τα λιγότερα χρήματα. Υπάρχουν κανόνες λοιπόν. Να σας υπενθυμίσω, ξέρω ότι όπως ξέρετε, διαφωνούσαμε για μήνες εδώ στην Επιτροπή για το πώς θα κατηγοριοποιήσουμε τις περιφέρειες. Είπαμε, επειδή το ΑΕΠ είναι το μόνο κριτήριο το οποίο ουσιαστικά σε όλη την Ευρώπη μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες τις περιφέρειες με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να το αξιοποιήσουμε ως το μόνο κριτήριο για μία πρώτη κατηγοριοποίηση. Μετά τα κράτη-μέλη μπορούν να κάνουν περαιτέρω διαφοροποίηση και μπορούν τους άλλους να μεταφέρουν πιστώσεις από τη μία περιφέρεια στην άλλη της χώρας τους. Αυτό υπάρχει στο γενικό κανονισμό. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν καλοί λόγοι που εφαρμόσαμε αυτούς τους κανόνες. Και μπορεί να φυγεί η Α ή η Β περιφέρεια και η δική μου περιφέρεια. Δεν έχουμε καμία δυνατότητα ε, να έχουμε ε, ενέργειες για την ενέργεια στη λειψεία που θα μας δημιουργούσαν θέσεις εργασίας. Ξέρουμε ότι οι δείκτες που χρησιμοποιούμε δεν μπορούν πάντα να είναι ο βέλτιστος τρόπος καθορισμού των πάντων αλλά είναι τελικά ο καλύτερος. Ξέρω ποια είναι τα προβλήματα των νησιών, δεν ήθελα να εμπλακώ στην συζήτηση για τα νησιά, αλλά ότι το κριτήριο ΑΕΠ είναι καλό και γι' αυτό το καθορίσαμε, αυτό ήθελα να αναφέρω. Για να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις και λάθος αντίπαλοι. Θέλετε να μιλήσετε εσείς ή η Επιτροπή. Λοιπόν, είχαμε διαπραγματική εντολή σαφέστατη. Αλλά παρακαλώ, να καταλάβετε ότι βασιζόταν στο ΝΑΤΣ 2, δηλαδή στο ΕΠ. Και η πρόταση ήταν όλα τα νησιά που είναι ΝΑΤΣ 2 να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο. Το κριτήριο δηλαδή το 75% του ΑΕΠ κατά κεφαλήν είναι, εφαρμόζεται σε επίπεδο ΝΑΤΣ 2. Συζητούσαμε λοιπόν τα νησιά ΝΑΤΣ 2 και χρησιμοποίησαμε το αντικειμενικό κριτήριο 75%. Όλα τα νησιά που αναφέρονται εδώ είναι πάνω από το 75%. Σαρδινία, Κορσική, Βαλιαρίδες και πώς θα λένε το άλλο. Αυτό ναι. Ευχαριστώ έχουν πάνω από 75% του ΑΕΠ κατά κεφαλή. Αν θέλετε μπορούμε να συζητήσουμε να περάσουμε σε ΝΑΤΣ 3, ΝΑΤΣ 4. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στο επίπεδο ΝΑΤΣ 2. Με βάση το ΝΑΤΣ 2 είναι πιο ανεπτυγμένες περιοχές. Προσπαθούσαμε να επιτύχουμε εξαιρέσει. Αν και γνωρίζουμε ότι είναι πάνω από 75% ας τις αντιμετωπίσουμε σαν να ήσαν λιγότερο ανεπτυγμένες. Σαν να είχαν κάτω από 75% αλλά η Κομισιόν ήταν κατά με βάση τη δική τους πείρα και ελπίζω το, η Κομισιόν τώρα να ε, μας το εξηγήσει. Το Συμβούλιο δεν είπε λέξη. Λέξη για τα νησιά. Εμείς υπερασπιζόμασταν τα νησιά, η Επιτροπή ήταν κατά, το Συμβούλιο μούγκα. Και εκεί καταλήξαμε. Είναι αντικειμενικό κριτήριο επίπεδο ΝΑΤΣ 2 που είναι ε, ε, ε, δείκτης εφαρμογής του Ταμείου Συνοχής. Και ξέρουμε ότι οι υπεραιτέρω δείκτες βασίζονται σε εθνικό επίπεδο. Τα νησιά αυτά λοιπόν κατέληξαν εκεί με βάση το εθνικό επίπεδο. Με το αντικειμενικό κριτήριο εξαιρέθηκαν τα νησιά αυτά. Επίσης εξετάσαμε εάν είναι εξόχως απομακρυσμένα τότε με βάση τη συνθήκη υπάρχει ειδική μεταχείριση. Χάσαμε, ναι. Αλλά χάσαμε αξιοποιώντα αντικειμενικά κριτήρια. Όχι υποκειμενικά. Αλλά παρακαλώ ρωτήστε τις κυβερνήσεις σας. Γιατί τα κράτη-μέλη δεν υπερασπίστηκαν τις περιοχές τους. Γιατί το Συμβούλιο δεν μας υποστήριξε. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Βεβαίω, υπάρχει ένα μείγμα κριτηρίων. Ο καθένας μας ξέρει την κατάσταση στη χώρα του. Στην ε, Πολωνία η περιοχή της ε, Βαρσοβίας είναι πλουσιότερη περιοχή, στις πλουσιότερες περιοχές λόγω της πόλης Βαρσοβίας, ενώ τα περίχωρα είναι ελάχιστα ανεπτυγμένα. Να ένα παράδειγμα. Ο συμβιβασμός λοιπόν βασίστηκε σε αντικειμενικό κριτήριο. Αλλά η Κομισιόν μας είπε ότι με βάση την πείρα της δεν θα έπρεπε τα νησιά επίπεδου ΝΑΤΣ 2 να τύχουν ειδική μεταχείριση. Γιατί δεν είναι εξόχως απομακρυσμένα. Και στατιστικά είναι πλουσιότερα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Το αποτέλεσμα είναι ένας συμβασμός. Πίτερ, να πεις εσύ, δύο λόγια. Έχουμε μακρηγορήσει, αλλά έτσι και αλλιώ προβλέπετε. Νομίζω ότι το βασικό είναι ότι εμείς δεν συζητάμε για ποσά. Μιλάμε για τον μηχανισμό ε, που θα επιτρέψει τη θεματολογική συγκέντρωση. Το θέμα των πιστώσεων είναι ένα διαφορετικό θέμα, είναι μια διαφορετική συζήτηση. Το θέμα είναι σε ποια επίπεδα θα, πρέπει να παραμείνουμε θεματολογική συγκέντρωση. Αυτό είναι το, το βασικό θέμα. Δεύτερον, η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι αυτού του τύπου ο μηχανισμός ε, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα εύχριστο, γιατί πιστεύουμε ότι ο πραγματικός τρόπος με τον οποίο θα πετύχουμε την εδαφική ολοκλήρωση είναι ακριβώς στην περιφερειακή ολοκλήρωση, είναι μέσω των προσπαθειών των, κρατήκων, των, των κρατών μελών, μέσω των δικών τους πολιτικών. Δεν κάνω τη διάκριση εγώ ανάμεσα στα νησιά ή στα βουνά. Το θέμα δεν μπορεί, δεν μπορεί να λυθεί με νομοθετικές ρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν οι από μακρισμένες περιοχές, έτσι και αλλιώς αυτό το κατανοούμε. Αλλά θέλουμε κάποιους γενικούς κανόνες που να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. Και γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι η προσπάθεια θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια του προγραμματισμού. Υπάρχει ένας μηχανισμός αντιστάθμισης, υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος προβλέπει ότι οι απαιτήσει συγκέντρωση μπορεί να μειωθούν στις ιδιαίτερα αναπτυγμένες περιοχές και το αντίθετο στις λιγότερο αναπτυγμένες. Όμως, ήταν ξεκάθαρο στα πλαίσια της συζήτησης και του τριμερούς διαλόγου ότι έπρεπε να βρεθεί μια κάποια λύση. Και αν πράγματι πρέπει να υπάρξει ένας τέτοιο μηχανισμός, απαιτούνται ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε εκ των υστέρων το τι έχουμε κάνει. Εξ αυτού λοιπόν, η διαδικασία πράγματι είναι μια διαδικασία συν Έγινε συζήτηση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και εμεί είχαμε τη θέση μας, αλλά το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είναι αυτοί που βρήκαν μια λύση. Και ένα επιπλέον σημείο σχετικά με τις ορεινές περιοχές, ορεινές ζώνες. Από ό,τι γνωρίζω υπάρχει μία πολιτική η οποία έχει ειδικού στόχους για τις ορεινές περιοχές, η ΚΑΠ, η οποία δεν είναι δική μας αρμοδιότητα και δεν είναι αρμοδιότητα του συγκεκριμένου επιτόπου. Ευχαριστώ Γιάνν. Θέλεις να δώσεις μια γενική απάντηση ή εντάξει, τέλειωσες με τα σχολιά σου. Νομίζω ότι οι παρατηρήσεις που έγιναν ήταν θετικές για τις ε, διαπραγματεύσεις, εκτός από τη συγκεκριμένη περίπτωση όπου δεν μπορέσαμε να εφαρμόσουμε πλήρως την εντολή που είχαμε. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συγγνώμη, στοιχεία ήταν ο μηχανισμός αντιστάθμισης. Εμείς συζητάμε το θέμα της θεματολογικής συγκέντρωσης εδώ και πάρα πολύ καιρό και στο τέλος έχετε κάτι που αλλάζει τα πάντα. Μία φράση. Τα κράτη-μέλη κάνουν ό,τι θέλουν καθορίζουν τα δικά τους όρια, τα δικά τους ποσοστά. Και σχετικά με τα νησιά είπαμε ότι τα πάντα μπορούν να κάνουν και να διορθώσουν τα κράτη-μέλη. Αυτή λοιπόν είναι η λύση στην οποία μπορούμε να καταλήξουμε. Τώρα, ε, αυτό ήταν μια μικρή φράση η οποία δεν υπήρχε στο αρχικό κείμενο. Ήταν κάτι το οποίο εισήχθη στο κείμενο μετά τις διαπραγματεύσεις. Είναι κάτι το οποίο καθιστά το συνολικό σύστημα ιδιαίτερα ευέλικτο. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώνουμε με το θέμα αυτό. Περνάμε τώρα στην εδαφική συνεργασία. Παρακαλώ τις ε, προτάσεις της έκθεσης αφήστε τες εδώ. Θα τα συλλέξουμε όλα εδώ και θα τα χρησιμοποιήσουμε εκ νέου. Ή αλλιώς πάρτε τα και φέρτε τα μαζί σας ε, την πρόταση έκθεσης τον ε, Ιούλιο γιατί δεν έχει νόημα να τα ξανατυπώνουμε. Περνάμε τώρα στο θέμα της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Πρόκειται για το σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Η κυρία Ρίκα Πακαρίναν δεν είναι μέλος μας πλέον. Και γι' αυτό θα ήθελα να αναφερθώ εγώ στα επιτεύγματά της, στα πλαίσια αυτής της διοργανικής διαπραγμάτευσης και μετά θα ζητήσω από τους Κιώδης και ιδιαίτερα από τη Μαρή να συμπληρώσουν τα λεγόμενά μου. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μετά τις διαπραγματεύσεις καταλήγουμε στη συνέχιση του ισχύοντος συστήματος με τα τρία επίπεδα συνεργασίας, δηλαδή διαμεθοριακή, ε, υπερεθνική και περιφερειακή συνεργασία. Γνωρίζουμε ακριβώς πώς λειτουργεί το Interreg και πώς ε, θα υπάρχει μια δυνατότητα συντονισμένη συνεργασία όλων αυτών των πολιτικών. Δεν έχουμε καταφέρει στο συγκεκριμένο τομέα εμείς να επιβάλλουμε μέσω των διαπραγματεύσεων για τις πολιετής προοπτικές αυξήσεις αυτές του 7% που επιθυμούσαμε. Εγώ ζήτησα από την ομάδα διαπραγμάτευσης και από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου να θέσουν το θέμα του ETC και του 7%. Αυτή ήταν η εντολή την οποία είχαμε σχετικά με το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, αλλά ε, σχετικά με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Εμείς προσπαθήσαμε στο εσωτερικό των ε, ε, υπαρχουσών πιστώσεων να μεταφέρουμε πιστώσεις προς την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, αλλά δεν πετύχαμε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Οπότε παραμένουμε στις αρχικές προτάσεις του Συμβουλίου στις πολιτικές αποφάσεις που είχε διατυπώσει το μήνα Φεβρουάριο σχετικά με τις ε, επενδυτικές προτεραιότητες και τη θεματολογική ε, συγκέντρωση. Νομίζω ότι σε σχέση με τους στόχους που είχαμε θέσει πετύχαμε κάποια πράγματα. Έχουμε πιο συγκεκριμένα ε, προγράμματα στόχους σε σχέση με τις αρχικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ζητούσαν μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερη υψηλότερη θεματολογική συγκέντρωση το 20% σαν παράδειγμα των διαθεσίμων πιστώσεων θα είναι απόλυτα δεκτικές σε κάθε ε, τύπο επένδυσης και το 80% θα ακολουθούν τέσσερους συγκεκριμένους στόχους. Θα υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο στοχολόγιο τετραπλό. Υπάρχει η δυνατότητα εδώ το 50% να ανταλλάσσεται ανάμεσα σε μεταφορές ανάμεσα στην διαμεθοριακή συνεργασία και στη διαπεριφερειακή συνεργασία και σχετικά επίσης με τις επενδυτικές προτεραιότητες καταφέραμε να βελτιώσουμε τη διατύπωση σε σχέση με την κινητικότητα των εργαζομένων, σε σχέση με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη βελτίωση της διαχειριστικής ικανότητας των δημοσίων υπηρεσιών. Είμαστε και πιο συμβατοί με τις προτεραιότητες ε, οι οποίες καλύπτονται και από τα Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Υπάρχει δηλαδή μεγαλύτερη συνέργεια ανάμεσα στους δύο διαφορετικούς κανονισμούς σχετικά με τον προγραμματισμό. Υπάρχει εδώ μια καλύτερη ευθυγράμμιση θα έλεγα της αρχικής πρότασης, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές. Και αυτό το οποίο πετύχαμε είναι η δυνατότητα να κρατήσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά που έχει αυτή η μορφή συνεργασίας και σε σχέση με την τεχνική βοήθεια, τεχνική αρρωγή και σε σχέση με συγκεκριμένους στόχους ανάπτυξης μέσω της συνεργασίας με τις λεγόμενες χώρες ΣΕΝΤ. Ε, which is, I think, important, which will be applied to all ε, programs, ε, is the, joint action plans επίσης έχουμε προχωρήσει ιδιαίτερα και στον τομέα της ολοκληρωμένης περιφερειακής ανάπτυξης και ανάπτυξης της υπαίθρου. Έχουμε καταφέρει να εισάγουμε στο σύνολο του συστήματος και κάποιες νέες μορφές εδαφικής συνεργασίας. μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στρατηγικές θαλασσίων λεκανών. Θα πρέπει επίσης να πω ότι γενικά πετύχαμε σαν διαπραγματευτική ομάδα. Στέφθηκε η προσπάθεια με επιτυχία. Θα πρέπει να προσθεθούν επίσης κάποιοι επιπλέον κανόνες ε, για τη συνεργασία ανάμεσα στις χώρες αυτές στο επίπεδο των ε, εξόχως μεμακρυσμένων περιοχών. Δεν μιλάω για δείκτες εδώ, ο Γιάνν δεν αναφέρθηκε σε δείκτες, εδώ μιλάμε για την εφαρμογή των οριζόντιων λεγόμενων κανόνων. Τα έχουμε ήδη συζητήσει αυτά. Αυτό το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο, και αυτό το διαπιστώνουμε οι συνάδελφοι που συμμετείχαμε στη διαπραγμάτευση, ήταν το θέμα και οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή τρίτων χωρών. Into account also the rules of the other funds which are involved in the cooperation when we talk about the cooperation. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα χαρακτηρίσει ε, τη συνεργασία μας με τις τρίτες χώρες. Το θέμα της απόστασης της ελάχιστης 150 χιλιόμετρων σαν παράδειγμα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για ορισμένες περιοχές, για όλους μας. Καταφέραμε επίσης στα πλαίσια της κακοφόρας συνεργασίας ανάμεσα σε όλα τα όργανα για το συγκεκριμένο θέμα, να εισάγουμε και πολύ μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή των κανόνων στους οποίους αναφέρθηκα την δυνατότητα μετά από αίτημα του συγκεκριμένου κράτους μέλους να προσθέσουμε κάποιες όμορες περιοχές στην εφαρμογή του προγράμματος. Δηλαδή υπάρχουν περιφέρειες ΝΑΤΣ 3 σαν παράδειγμα οι οποίες θα μπορέσουν να διευρυνθούν, θα μπορέσουν να συμπεριλάβουν και να συμπεριληφθούν και επιπλέον περιφέρειες. Και υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και σε σχέση με τη την ε, θεματολογία των περιοχών τρίτης κατηγορίας. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εξ ναι. ονόματος ε, της ΡΙΙΚΑ, παρά λοιπόν το ότι, ότι χάσαμε το 7%, νομίζω ότι κατά τα άλλα η διαδικασία ήταν κερδοφόρα. Η Μαρή Τερέζ θα με συμπληρώσει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να χαιρετήσω την πρώτα των συζητήσεων που είχαμε στον τριμερή διάλογο. Ήταν τεχνικά ενδεχομένω ενίοτε τα θέματα και ενδεχομένω και δύσκολα για πολλού να τα παρακολουθήσουν, πολύπλοκα, αλλά τελικά το Κοινοβούλιο πέτυχε. Όχι βέβαια εφόλων των σημείων, αλλά πετύχαμε πρόοδο. Αυτό είναι και η πρόκληση στις ε, διοργανικές διαπραγματεύσεις. Αναγκαστήκαμε και εμείς να κάνουμε συμβιβασμούς, εγκαταλείψαμε κάποια σημεία και κερδίσαμε σε κάποια άλλα είναι οι κανόνες του παιχνιδιού. Σε ό,τι αφορά το, τα πολλά και διαφορετικά έγγραφα τα οποία λαμβάναμε και την τελευταία στιγμή πολλές φορές, ε, τεράστια, ε, τεράστιους όγκους χαρτιών συγκεντρώσαμε που δεν ήταν και πάντα επικαιροποιημένα. Τέλο πάντων μας δυσκόλεψε όλο αυτό. Χρειάστηκε επίσης να συντονιστούμε και με τους άλλους κανονισμούς που συζητούν στο πλαίσιο άλλων τριμερών διαλόγων και δεν συμμετέχουν όλοι βουλευτές σε όλους τους τριμερείς διαλόγους. Ήταν δύσκολος ο συνδυασμός σε κάποιες φορές. Σε ό,τι αφορά τώρα του θεματικού στόχου, τέθηκε το θέμα, αναφέρθηκε επενδυτικέ προτεραιότητε ε, στο πλαίσιο τη συνολική συνεργασία. Η πρόταση τη Κομισιόν, η οποία πρόσθεσε κάποιε προτεραιότητε, ε, ειδικέ επενδύσει ε, για τον κανονισμό τη εδαφική συνεργασία. Τροποποίησαμε τι προτάσει αυτέ, προτείναμε και προσθέσαμε νέε. Κάτα τις διαπραγματεύσεις Πολλές από τις, από τις τροπολογίες μας έγιναν ε, αιτιολογικές σκέψεις, ε, διότι ήταν ε, ανάγκη να συμμορφωθούμε και με τις διαπραγματεύσεις ό,τι αφορά το ΕΤΠΑ. Κάποιες φορές αναφερόμαστε στο ΕΤΠΑ, κρατήσαμε κάποιες προτεραιότητες ως επιλογή και στις αιτιολογικές σκέψεις αναφερθήκαμε σε κάποιες άλλες να υπενθυμίσω κάποια επιτέγματα, όπως είπε και η πρόεδρος, να τα υπενθυμίσω και εγώ. Πρώτα απ' όλα, ε, επιλεξιμότητα των εξόχως προμακρυσμένων περιοχών για την ε, διασυνορική συνεργασία. Ε, με τον κανόνα αυτό των 150 χιλιόμετρων που περιορίζει ε, την απόσταση τη θαλάσσια συνεργασία. Το Συμβούλιο και η Κομισιόν ήταν ε, κάθετα αντίθετο με την ελάφρυνση του κανόνα. Εμείς επιμείναμε για την επιλεξιμότητα όταν ζητάει ένα κράτος μέλος και για τις εξόδους απομακρυσμένες περιοχές αλλά και για τα μικρά νησιά της ίδιας θαλάσσιας λεκάνης γίνεται. Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων πείσαμε με δυσκολία τα άλλα διαθεσμικά όργανα για να γίνουν επιλέξιμες και οι εξόχως απομακρυσμένες ε, περιοχές στο πλαίσιο της εθνικής επικράτειας του κράτους. Υπήρξε άρνηση όμως ε, μήπως ε, με το φόβο ότι μπορεί να είναι πάρα πολύ ε, ο κατάλογο των επιλέξιμων περιοχών και υπάρχει πρόβλημα με τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές και θα καταθέσουμε τρόπολογίε γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι επιλέξιμα κάποια νησιά. Ε, τα κράτη-μέλη ε, μπορεί να το επιθυμούν, άρα μπορούν κάτι να κάνουν, όπω είπε και ο εισηγητή. Ό,τι αφορά τις διασυνοριακέ επενδύσεις διατηρήθηκε το, το ΕΤΠΑ, το ΠΙΣ το 80% έχουμε στους τέσσερις στόχους και 20% ελεύθερο στο πλαίσιο θεματικής συγκέντρωσης, πιστοποίηση για να έχουμε παρακολούθηση και ε, της, ε, των πληρωμών, ε, προσαρμογή των μικρών προγραμμάτων και κάποιες επενδυτικές προτεραιότητες συγκεκριμένε για τα προγράμματα ανταλλαγής καλών πρακτικών Interactor Back Το πιο μεγάλο πρόβλημα βέβαια αναφέρθηκε, κοινοπροϋπολογισμός... Η κυρία Πρόεδρος είπε ότι είχαμε στήσει 7%, η Κομισιόν πρότεινε 3,4% και 2,7% νομίζω το Συμβούλιο. Δεν είναι αποδεκτό αυτό από εμάς. Δυστυχώς επίσης εγκαταλείψαμε και ήταν πολύ προσφυλές για μένα ε, της, την κατανομή άνα πρόγραμμα. Θα γίνει μια μελέτη από την Κομισιόν για τη σκοπιμότητα ε, να υιοθετηθεί τέτοιο μέτρο στο μέλλον. Ζητήσαμε σε αντάλλαγμα να αυξηθεί, μάλλον να δοθεί ε, κονδύλι μεγαλύτερο για την αδαφική συνεργασία. Και θα πρέπει να κάνει μια νέα κατανομή η Κομισιόν, δεν ξέρω αν την έχει ήδη ολοκληρώσει. Τέλος, ε, μια τελική σκέψη ζητάμε αν μπορούν οι περιφέρειές μας συνεργάζονται με περιφέρειες τρίτων χωρών στο πλαίσιο της ε, διαπεριφερειακής συνεργασίας που ήδη είναι δυνατή σήμερα και γνωρίζω ότι ο συνάδελφο ε, Όλμπριχτ και ο συνάδελφο Φανή Τελερό δραστηριοποιούνται ενεργά στον τομέα αυτό. Το Συμβούλιο όμω μπλοκάρει την κατάσταση, είναι διχασμένη η Κομισιόν. Θα επανακαταθέσουμε αύριο αυτή την τροπολογία, ελπίζω να τύχει τη υποστήριξή σα και τέλο θέλω ε, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την ε, Ρίκα για την δουλειά της και για το ευτυχές γεγονός που αναμένει να τις ευχηθούμε, να τις στείλουμε να Ευχαριστώ. Thank you, Marie Σας ευχαριστώ Μαρή Φραντσέσκο δεν είναι εδώ. Ο Φρανσό Αλφονζή λοιπόν. Κυρία Πρόεδρο, όπως συμπλήρωσε και η είχε θετικά αυτή η διαπραγμάτευση. Βελτιώθηκε ο κανονισμό, συμπεριλήφθησαν ορισμένα θέματα που ήθελε να προωθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εδαφική συνεργασία. Ωστόσο, Νομίζω ότι η ανάπτυξη εδαφικής συνεργασίας είναι μεγάλη φιλοδοξία του Κοινοβουλίου και τη Επιτροπής και για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού 14-20. Ε, η οικονομική όμως αντιμετώπιση το Φεβρουάριο με τις διαπραγματεύσεις των Βρυξελών ήταν καταστροφική. Δηλαδή έχουμε πλέον προϋπολογισμούς που δεν θα είναι μεγαλύτεροι σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Έχουμε ε, τις μακροστρατη... μακροπεριφικές στρατηγικές και πολλά άλλα εργαλεία για να αναπτύξουμε αυτή την πολιτική που είναι μια μείζον ευρωπαϊκή πολιτική εξορισμού. Λοιπόν, πραγματικά που βλέπω σε ποιο βαθμό το Συμβούλιο, τα κράτη επέδειξαν ελάχιστη φιλοδοξία για την αδαφική συνεργασία. Αν είναι δυνατόν και την αδαφική συνοχή, αν μπορούμε ε, να δώσουμε μεγαλύτερο εύρος σε αυτή την πολιτική. Αν έχουμε κάποια περιθώρια πρέπει να το πράξουμε. Πρόεδρος, πριν δώσω το λόγο σε άλλους συναντέλφους, θα ήθελα να πω κάτι που το ξέχασα, αλλά είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου. Δηλαδή ότι για πρώτη φορά έχουμε ένα ξεχωριστό ρυθμιστικό πλαίσιο για αυτή την πολιτική. Πρόεδρός ήταν αυτή που πρώτη το είπε στη Λέγη Επιβελικής Προεδρίας. Τότε για πρώτη φορά το είπαμε φωναχτά, δεν υπήρχε συμφωνία τότε στο Συμβούλιο για χωριστό κανονισμό. Στηρίξαμε τις προσπάσεις Κομισιόν να προχωρήσουμε με ένα ξεχωριστό κανονισμό και έτσι έχουμε αυτή την πολιτική, την ολοκληρωμένη, την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. Δεν σας βλέπω κυρία Κρέλ, κάντε εκεί πέρα καμία χειρονομία να σας βλέπω. Με συγχωρείτε, δεν κατάλαβα ότι πρέπει να είμαι σκιώδης και για αυτό το θέμα, γιατί ο Φραντσέσκο λείπει. Θα σας το διαβάσω. Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για την εργασία που έκανε η συγγήτρια και η πρόεδρος. Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων δείχνει ότι η στενή συνεργασία μεταξύ των διαπραγματευτών του Κοινοβουλίου είναι όχι μόνο επιθυμητή, αλλά υποχρεωτική για να επιτύχουμε σημαντικά αποτελέσματα. Από πλευρά πόρων πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει αύξηση για την εδαφική συνεργασία το 2,75% είναι απαράδεκτο. Πολύ κάτω από το 7% που είχε προτείνει το Κοινοβούλιο στο, στην εντολή της ΡΕΓΚΙ. Καλωσορίζουμε τις βελτιώσεις για περισσότερη τυποποίηση, απλοποίηση διαδικασιών με βάση τα αιτήματα του Κοινοβουλίου και την ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη που θα καλύψει και περιφέρειες στο ΝΑΤΣ 3, των οποίων τα θαλάσσια σύνορα ε, ε, ε, απέχουν τα μένα εκ των δε περισσότερο από 150 χιλιόμετρα. Επίσης περισσότερη ευληγησία για την επιλογή εταίρων και τις προτεραιότητες επενδύσεων βοηθούν τις τοπικές οργανώσεις και τις περιφέρειες για να υπάρξουν απλουστευμένες διαδικασίες για το στόχο που επιδιώκουμε. Οι διαδικασίες αυτές στο παρελθόν δεν ήταν έχουστες και ήταν περίπλοκες. Η άλλη σκιώδη λέει πρόεδρος δεν είναι εδώ. Οπότε ο Λαμπέρ Φανίστελρόι. Λοιπόν, υπάρχει χωριστός κανονισμός, αλλά έχουμε λιγότερε λιγότερες πιστώσεις. Εφού λοιπόν τώρα είναι χωριστό, δεν έχουμε δυνατότητες μεταφορών από άλλα σημεία. Ναι, μεν ε, χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτό που επιτύχαμε, αλλά είναι πολύ λυπηρό το αποτέλεσμα. Τι μπορεί να επιτύχει. Ανάμεσα σε αυτά που είχαμε και αυτό που έχουμε τώρα είναι απαράδεκτο. Η Πρόεδρος έστειλε ήδη μια επιστολή από πλευράς όλης της Επιτροπής για να ζητήσει περισσότερους πόρους. Ευκταίο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι ρεαλιστικό. Μετά χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό για να είναι πιο ευέλικτη η εφαρμογή. Ξέρετε τη συζήτηση που κάναμε στην αρχή της εξέτασης. Τότε είχαμε καταφέρει να δοθεί περισσότερη προτεραιότητα στην διαμεθοριακή συνεργασία. Είναι ενα από τους κύριους στόχους που επιτύχαμε. Θα πρέπει να βελτιωθεί η διαμεθοριακή συνεργασία. διότι το 2,75% είναι υποχώρηση. Ας δούμε όλοι μαζί, σκιώδεις, συνάδελφοι, πώς μπορούμε ε, να επιτύχουμε περισσότερη ευελιξία χρειαζόμαστε ε, διάφορου εταίρου από διάφορε χώρε σε αυτή τη διαμεθοριακή συνεργασία και ναι, μεν μπορούν να το κάνουν οι χώρε, αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουν όλε. Ευχαριστώ. Η Ρώσα. Ευχαριστώ. Αυτό για τα 150 χιλιόμετρα. Μιλάγαμε προηγουμένως για αντικειμενικά κριτήρια. Γιατί 150 και όχι 200 ή 250. Εγώ ρώτησα τον Επίτροπο ποιο είναι το κριτήριο και μας είπαν ότι επειδή αυτό το πρόγραμμα ξεκίνησε από τα νησιά της Βαλτικής βάλανε 150 χιλιόμετρα τότε. Θα μπορούσαν να βάλει 200. Να αντικειμενικό κριτήριο. Όταν μας βολεύει το ΑΕΠ ε, βάζουμε το ΑΕΠ, όταν μας βολεύει η απόσταση βάζουμε την απόσταση. Οπότε σημαίνει ότι οι Βαλεαρίδες δεν θα έχουν ούτε θεματική συγκέντρωση, ούτε και δυνατότητα διαμεθορικής συνεργασίας. Για το ένα λόγο του ΑΕΠ και για το άλλο για λόγους απόστασης. Ενώ η συνθήκη λέει ότι πρέπει να ε, δοθούν περισσότερες δυνατότητες να αποκατασταθεί το μειονέκτημα, να αντιμετωπιστεί το μειονέκτημα των νησιών. Και δεν αποκαθίσταται τίποτα. Η συνθήκη δεν λέει ε, ότι πρέπει να ε, αποζημιωθούν τα νησιά λόγω του μειονεκτήματός τους, λέει μόνο αυτό, δεν μιλάει για ΑΕΠ. Οποιοδήποτε νησί έχει προβλήματα στην εκπαίδευση, στις μεταφορές, στη βιομηχανία, στη γεωργία, στην υγεία. Ξέρετε ότι είναι τέσσερα τα νησιά των Βαλεαρίδων που ξέρω καλύτερα που είναι άνισα και μεταξύ τους. Τα κριτήρια λοιπόν είναι μια έτσι, μια αλλιώ. Με συγχωρείτε, εγώ διαφέρω, διαφωνώ. Θα συνεχίσω να ε, ζητάω την κατάργηση των 150 χιλιόμετρων για να μπορούν να έχουν και οι βαλερίδες πρόσβαση σε αυτούς τους, ε, σε αυτούς τους πόρους. Ο Μποστινάρου για το Ταμείο συνεχίζω. Ευχαριστώ. Όπως ε, και σε προηγούμενες ενημερώσεις τονίζω ότι επιτύχαμε να διατηρήσουμε, να προστατεύσουμε και εν τέλει να επιτύχουμε πλήρως τους στόχους μας. Επιτύχαμε λοιπόν το στόχο μας. Αποστολή εξετελέστη. Όπως λέγεται σε πολλές γλώσσες. Λοιπόν, θα είμαι κατά τα υπόλοιπα επιγραμματικός. Ορισμένα σημεία δεν έχουν κλείσει ακόμη. Θα κλείσουν μέσω τροπολογιών που θα υποβάλουμε στην έκθεση, ανάλογα και με άλλες εξελίξεις. Ένα αφορά το 2 bis για το Ταμείο Συνοχής, ενίσχυση του μέσου συνδέοντας την Ευρώπη. Αυτό είχε μπει στο πεδίο ε, εφαρμογής του Ταμείου Συνοχής, ενώ τώρα είπαμε να μπει σε άλλο άρθρο. Το περιεχόμενο δεν διαφέρει από την άποψη του Κοινοβουλίου, από τη θέση του Κοινοβουλίου θα αναφερθεί ότι το Ταμείο Συνοχής θα υποστηρίξει προγράμματα υποδομής εντός του μέσου συνδέοντας την Ευρώπη με βάση του άρθρου 84% του CPR όπου θα περιλαμβάνεται η συμφωνία που επιτύχαμε και που εγκρίθηκε και από τη Ρέτζη και από την Τραν και που θα τον αναλάβει η Γενική Διεύθυνση MOVE. Ένα νομικό θέμα, αλλά σημαντικό. Το Ταμείο Συνοχής δεν δημιουργήθηκε μέσω της συνθήκης. Η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου διερευνά, διερευνούν μία νομική λύση για το θέμα αυτό για να μην υπάρξει καμία νομική αβεβαιότητα. Θα περιμένουμε την άποψή τους. Θα αλλάξουν κάπως οι αιτιολογικές σκέψεις για να αντανακλούν αλλαγές στα άρθρα. Θέλουμε επίσης να διατηρηθεί το αιτιολογικό, ε, η αιτιολογική σκέψη που ε, αναγράφει την αρχή «Ο Μολύνων πληρώνει» που εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή μας. Και η Κομισιόν ήταν υπέρ, αλλά η Προεδρία ακόμη ε, αντιτίθεται. Ψάχνουμε μια λύση. Τι επέτυχε λοιπόν αυτή η έκθεση. Ενεργειακή αποτελεσματικότητα και ανανεώσιμες για προγράμματα ε, ιδιωτικών κατοικιών ενώ η πρότασή μας μιλούσε μόνο για δημόσια κτίρια συμπαραγωγή και υψηλής ε, απόδοσης θέρμανση, επενδύσεις για την ίδρυυση και την αποχέτευση μεγάλης κλίμακας, οικοφιλικές μεταφορές και επιτύχαμε μεγάλο ποσοστό συντονισμού με το ΕΤΠΑ για να υπάρχουν σαφέστερες διατάξεις και ευχερέστερη εφαρμογή. Θέλουμε ταυτόσιμες διατάξεις για ταυτόσιμους επενδυτικούς στόχους. Δεν έχει υπάρξει, αποφάσεις, δεν έχει υπάρξει απόφαση για την μακροοικονομική αιρεσιμότητα και είπαμε ότι θα το αφήσουμε αυτό στο CPR. Θα το αφήσουμε λοιπόν στην Επιτροπή ε, Περιφερειακής Πολιτικής και θα, ε, εφόσον υπάρξει συμφωνία, θα μπει στον κανονισμό του Ταμείου. Για τους κοινού δείκτες, ίδιοι κανόνες με το Ταμείο Συνοχής, ίδια διατύπωση. Ταυτόσημη. Ευχαριστώ λοιπόν τους πάντες και ενημερώνω ότι ε, μέχρι αύριο το μεσημέρι είναι η προθεσμία υποβολή τροπολογιών. Αλλά λόγω τη θαυμάσια συνεργασία με όλου του σκιώδει, με όλου του συναδέλφου και με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, θεωρώ ότι δεν θα χρειαστούν τροπολογίες ούτως ώστε η έκθεση που είναι το αντικείμενο διαπραγμάτευσης τους τριμερείς διαλόγους να μπορέσει να ψηφιστεί στην ε, Ρέτζη τον Ιούλιο χωρίς ε, αλλαγές. Υπογραμμίζω και πάλι ότι στο κανονισμό για το Ταμείο Συνοχής η Επιτροπή ήταν ευέλικτη, έδειξε πολύ θετικό πνεύμα συνεργασίας και συνεργάστηκε με το Κοινοβούλιο για να εξευρεθούν οι βέλτιστες λύσεις και επειδή συνεργαστήκαμε καταφέραμε να πείσουμε και το Συμβούλιο στην αρχή των ε, συζητήσεων δεν ήταν προφανές ότι θα μπορούσαμε να επιτύχουμε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ την Κομισιόν και προσωπικά τον Πίτερ Μπέρκοβιτ. Εγώ ελέγχω εδώ την πρόταση εκθέσης και δεν βλέπω την κατάργηση της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας. Θα το ελέγξουμε, ίσως να υπάρξει να χρειαστεί ένα διορθωτικό. Γιατί ξέρετε ότι το διαγράψαμε από την πρόταση. Τελειώσαμε λοιπόν. προλαβαίνουμε να κάνουμε τον Ιακίμ τώρα. Όχι. Μετά τον Βίκτορ θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Οι σκιώδεις δεν είναι παρόντες. Έχουν φύγει. Δεν υπάρχει κάποιος που θα πάρει το λόγο για την έκθεση του Βίκτορ. Λοιπόν, ή τελειώνουμε με αυτό ή κάνουμε την έκθεση του Ιωακίμ. Πιστεύετε ότι μέσα σε 10-15 λεπτά και αύριο τότε θα αρχίσουμε λίγο αργότερα. Τσέλερ. Ευχαριστώ. Επανειλημμένα έχουμε συζητήσει για την τροποποίηση του κανονισμού αυτού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας. Ε, είχαμε επιτύχει μια σημαντική πρόοδο. Αν δείτε το σχέδιο έκθεσης βλέπετε μόνο το άρθρο, όχι τις αιτιολογικές σκέψεις. Γιατί, επειδή ήθελα να δείξω καλή διάθεση. Πολλά τα, που ήθελα να είναι στο άρθρο, τα έβαλα στα άρθρα, τα έβαλα στα, ε, στις αιτιολογικές σκέψεις. Γιατί έτσι τουλάχιστον υπάρχουν μέσα στο κείμενο και μπορούν να αξιοποιηθούν μετά. Ε, αναφερόταν λοιπόν η ε, σιωπηρή ε, έγκριση και ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμπεριληφθούν όπως και δημόσιες, δημόσιοι οργανισμοί στην συνεργασία αυτή. Είχαμε μόνο τρεις επίσημες συναντήσεις, τριμερούς διαλόγου, αλλά είχαμε και διάφορες άτυπες συναντήσεις όπου ανταλλάξαμε απόψεις για να διευκρινιστούν τι εννοούσε ο καθένας, γιατί είναι πολύ τεχνικά αυτά τα θέματα. Και ε, νομίζω ότι όλοι και αυτοί που δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με αυτό το θέμα καταλαβαίνουν την σημασία του. Αυτό που πρέπει να διαπιστώσω είναι ότι ναι μεν εμείς νομίζουμε ότι επιτύχαμε συμφωνία, αλλά υπάρχουν ακόμη κάποιες ε, χώρες μέλη που θεωρούν ότι η δημιουργία αυτού του θεσμού είναι προσβολή της κυριαρχίας τους. Και θεωρούν ότι θα μπορούσαν να ξεφύγουν από τον έλεγχό τους αυτές οι ε, δραστηριότητες αυτών των οργανισμών, γιατί είναι ε, διαμεθοριακές αλλά υπήρχαν ούτως άλλως ε, προηγουμένως και τέτοιες οργανώσεις. Παρ' όλα αυτά ορισμένοι δεν θέλουν να κατανοήσουν γιατί πρέπει να υπάρχουν. Θέλουμε να ενισχύσουμε αυτή τη δυνατότητα για να προωθήσουμε την διαμεθοριακή και διεθνική συνεργασία και να την διευκολύνουμε. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε περαιτέρω δυσχέρειες. Αφού λοιπόν μετά συμφωνήσαμε, οι αιτιολογικές σκέψεις που ήταν περίπου 40 ε, επιχειρείται να τροποποιηθούν μέσω της γραπτής οδού και κυρίως μέσω της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου φαίνεται να θεωρείται ότι εγώ τους υπέβαλα ορισμένα πράγματα τα οποία δεν τα κατάλαβαν και τα οποία ε, μπορούν να είναι αντικείμενα παρερμηνιών. Εάν λοιπόν αυτά που είναι στις ε, αιτιολογικές σκέψεις δεν είναι σαφή, μπορούμε επίσης να ε, τα, τις συμπεριλάβουμε και σε περαιτέρω διακηρύξεις δικές μας εάν δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε τα πάντα. Αλλά ορισμένα πράγματα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. Τελειώ δεν χρειαζόμαστε καθόλου ένα νέο κανονισμό. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε να απαλληφθούν όλα. Ε, γιατί αλλιώ δεν θα χρειαζόταν λοιπόν να έχουμε κάνει όλη αυτή την προσπάθεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσω να συνοηθώ και αν δεν τα καταφέρουμε κατά την Ιρλανδική Προεδρία, τότε θα επιχειρήσω να συνοηθώ με τη Λιθουανική Προεδρία, γιατί επειδή έχουν ήδη υπάρξει προσδοκίες για αυτό το νέο κανονισμό και πολλοί με ρωτάνε πώς, πότε θα έχουμε αυτό το νέο κανονισμό που είναι πιο ευέλικτο και που επιτρέπει πιο ε, πλούσια και πιο διαφοροποιημένη εδαφική συνεργασία και γι' αυτό νομίζω ότι τελικά δεν θα καταφέρουν να μας σταματήσουν. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κανείς όδης εδώ. Δεν το βλέπω. Α, η Κωνσταντσε. Να σε καλά Κωνσταντσε. Κανείς άλλος θέλει να συζητήσει κάτι, να πει κάτι. Ο Γιώργη τα κατάφερε καταπληκτικά από ό,τι βλέπω εδώ. Ήταν πάρα πολύ μεγάλες οι τεχνικές και νομικές δυσκολίες. Αν και σύντομη εντόμη έκθεση άκρος δύσκολη. Ουδή θέλει το λόγο από ό,τι βλέπω. Α, Σον. Κέλλη, είναι προσωπικό το θέμα. Ουσιαστικά λόγω της εθνικότητάς μου, ο Γιώαχημ αναφέρθηκε στην Ιρλανδική Προεδρία δύο φορές. Και γνωρίζω ότι υπήρχαν ε, σε επίπεδο επιτροπής εδώ κάποια προβλήματα ότι δεν έχει γίνει επαρκής πρόοδος ε, από την Ιρλανδική Προεδρία υπήρχε, υπήρχαν κάποιες κριτικές, αναφερθήκατε και στις ε, πολυπλοκότητες και στις τεχνικές δυσκολίες. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να ανακύψει με την οποιαδήποτε προεδρία μέχρι ότου καταλάβει ε, όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με μια πρόταση. Νομίζω ότι τις διαπραγματεύσεις ε, τις προεδρεύσαμε επιτυχώς και προχωρήσαμε, σημειώσαμε πρόοδο. Ποια είναι τη δράση τώρα από τους συμμετέχοντες επί του διαλόγου. σε σχέση με τη συμμετοχή και την ε, προσήλωση της ε, Ιρλανδικής Προεδρίας στα θέματα που απασχολούν την ε, Περιφερική Επιτροπή. Νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν παράπονα. Ο, η Πρόεδρος, δεν υπάρχουν άλλοι που θα το δώσω στο Γιάχη. Λοιπόν, να απαντήσω σε αυτό που είπε ο κύριος Κέλλη. Αν άκουσες προσεκτικά, δεν επέκρινα την Ιρλανδική Προεδρία. Μπορώ να καταλάβω ότι οι διαπραγματευτές της Ιρλανδικής Προεδρίας για ένα τόσο δύσκολο νομικό και τεχνικό θέμα βεβαίως βασίζονται σε αυτά που τους λένε οι υπηρεσίες και τα κράτη-μέλη και αν έχουν διάθεση συνεργασίας. Και εκεί υπήρξαν αδυναμίες. Δεν υπήρχε η αναγκαία διάθεση συμβασμού από πλευράς κάποιων κρατών μελών, όπως φαίνεται και από διάφορα εσωτερικά έγγραφα που είδα. και επίσης υπήρξε και πρόβλημα κατανόησης. Αλλά αν κάποιοι δεν καταλαβαίνουν κάτι για κάποιο θέμα, δεν πρέπει να διαπραγματεύονται για αυτό το θέμα. Και ε, ε, ε, υποστηρίχθηκαν νομικές απόψεις οι οποίες λείπησαν ιδιαίτερα την Ελλαδική Προεδρία. Ωραία, λίγη συνεδρίαση. Επειδή έληξαν όλα τα θέματα που είχαμε μέχρι αύριο 10.30. Μπορούμε να συνεδριάσουμε στις 10.30, αλλά 10.30 θα αρχίσει η ψηφοφορία. Οπότε πρέπει στις 10.25 να είστε στην αίθουσα. Παρακαλώ να ενημερώσετε όλοι ότι θα αρχίσει η ψηφοφορία 10.30. Θα κυκλοφορήσει και η ενημέρωση. Λοιπόν, λίγη συνεδρίαση και έχουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών. Παρακαλώ.